των και θα αρχίσουμε σε λίγο τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καθίστε παρακαλώ για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Για να πάει κάποιος να ψάξει τον κύριο Μάντες, που είναι το πρώτο μας θέμα στην ημερήσια διάταξη. Είναι εδώ. Στο μεταξύ, σας καλωσορίζω όλους εδώ στην συνεδρίασή μας αυτή σήμερα το απόγευμα, σε αυτή τη σκοτεινή αίθουσα. Έχουμε και λίγο χώρο, δεν έχουμε και φω τη ημέρα, αλλά ήταν η μόνη ελεύθερη από ό,τι φαίνεται. Να ξέρετε επίση ότι περνά στον κυβερνοχώρο η συνεδρίαση αυτή. Και γι' αυτό και θέλω να ξεκινήσουμε στην ώρα μα γιατί κάποιο κάπου μπορεί να θέλει να μα παρακολουθήσει. Δεν μπορεί να καθυστερούμε. Πρώτα απ' όλα, ξεκινήσουμε με την έγκριση τη ημερήσια διάταξη. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Ωραία, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Τώρα, ανακοινώσει του Πρόεδρου. Θέλω να σας ανακοινώσω κάποιες αποφάσεις που πήραν οι συντονιστές πριν από λίγο. Πρώτα απ' όλα, ότι ορίσαμε εισηγητέ για ορισμένες εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας που αποφασίστηκαν από τη διάσκεψη των Προέδρων. Πρώτον, των μέλων της Ευρωπαϊκής Τυποποίησης, από την ομάδα των συντηρητικών, ο κ. Σίσκερ. Επίση, οι επιπτώσει τη διαφήμιση της συμπεριφορά των καταναλωτών, κάποιο από το ΕΛΚ θα το αναλάβει αυτό. Και για μια έκθεση όσον αφορά την οδηγία για την ασφάλεια και την εποπτεία της αγοράς που θα αναλάβει κάποιος από τους σοσιαλιστές. Όλες αυτές οι εκθέσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές είναι, βοηθούν στον νομοθετικό χαρακτήρα της Επιτροπής μας. Επίσης γνωμοδότηση για την Νομική Επιτροπή και η Επιτροπή Αναφορών επίσης μας μετέφερε μία αναφορά για να εξετάσουμε θέματα που έχουν να κάνουν με την εισαγωγή κρέατος καγκουρό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συντονιστές θα το δουν αυτό ξανά για να αποφασίσουν ποιος θα αναλάβει αυτό το θέμα. Θέλω πάντως να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Επιτροπής μας και τους συντονιστές ιδιαίτερα που βοήθησαν να πετύχει η συζήτηση keynote στο Στρασβούργο που είχαμε για τρεις ε, εκθέσεις πρωτοβουλίας, ε, Hunhead και Buzoi, για το βαθμολόγιο της εσωτερικής αγοράς, όπως επίσης και τη στρατηγική Solvit. Νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερα επιτυχής οι συζητήσεις μας αυτές. Τώρα, οι συντονιστές επίσης ενέκριναν, συμφώνησαν μάλλον, για ένα πρόγραμμα εργασίας όσον αφορά την αποστολή μας στην Ελβετία, όσον αφορά τις εξωτερικές δραστηριότητές μας. Τέλη Μαΐου λοιπόν η Επιτροπή μας θα πάει σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς ε, της για παράδειγμα, για να προετοιμάσουμε τις δικές μας εκθέσεις πρωτοβουλίες για την τυποποίηση όπως σας είπα πριν. Και επίσης θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια νέα διαδικασία προκειμένου η Επιτροπή να προβαίνει σε διαθρωμένο διάλογο με αρμόδιους επιτρόπους για το νομοθετικό πρόγραμμα 2010 και 2011. Φροντίζουμε λοιπόν γι' αυτό και θα σας αρέσει να ακούσετε ότι έχουμε περιορισμένο αριθμό μεγάλων προτεραιοτήτων ως Επιτροπή που πρέπει να εγκρίνουμε και ίσως να εντοπίσουμε και κάποιες αρνητικές προτεραιότητες. Έτσι λέει. Ε? Που δεν θέλουμε δηλαδή να συμπεριλάβουμε. Καταλαβαίνετε πόσο ενδιαφέρον θα είναι ο διάλογος αυτός με τους επιτρόπους για τις αρνητικές μας προτεραιότητες. Αυτός είναι ο όρος. Οι συντονιστές λοιπόν θα κοιτάξουν τι ομάδες εργασίες, τι μελέτες μπορούν να γίνουν ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα περί 2020. Τώρα όμω έρχομαι στον εισηγητή μας τον κύριο Μάντερς που έχει μια πολύ σημαντική έκθεση για ονομασίε και συναφείς επισήμανση κλωστοϊφαντουργικών προϊόντων. Έχουμε εδώ και σκιώδεις εισηγητές, Κόμες, Αρντεμόσα, Ρούλε Μακλάκεν και Σβένσον. Α, δεν είναι εδώ. δίνει. Κύριε Μάντερς, παρακαλώ, έχετε το λόγο για να μας παρουσιάσετε την κατάσταση πραγμάτων όσον αφορά την έκθεσή σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι έχετε όλο το σχέδιο εκθεσής μου. Θέλω να ευχαριστήσω τους κοιόδες εισηγητές ευθύς εξ αρχής για την καλή συνεργασία που είχαμε μεταξύ μας. Είναι πολύ ωραίο να βλέπει κανείς τι ωραία που μπορούμε να συνεργαζόμαστε και ότι έχουμε τις ίδιες απόψεις όσον αφορά το μέλλον της επισήμασης κλωστοεφαντουργικών προϊόντων. Την προηγούμενη φορά είχα κάτι σπορ παπούτσια μαζί μου, τώρα έχω κάτι άλλο μαζί μου και είναι για να σας δείξω τη σήμανση στα προϊόντα αυτά. Να, κοιτάξτε. Μπορώ να το δώσω να γυρίσει στην αίθουσα να το δείτε. Υπάρχουν εδώ πέρα τέσσερα κομματάκια. Ε, υφάσματα βλέπετε. Γι' αυτό το πράγμα. Καλά, δεν είναι για να γελιοποιήσουμε το θέμα, όχι. Αλλά είναι για να σας εξηγήσω ότι πώς είναι δυνατόν να βάλουμε 22 γλώσσες εδώ μέσα. Στο σχέδιο εκθεσής μου ζητάω από την Επιτροπή Ξέρω ότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε στάνταρ μεγέθη, μόνο μία γλώσσα, η σύμβολα κτλ. Όχι, χρειάζεται πρώτα έκθεση εξολόγησης για κάτι τέτοιο. Αυτό λοιπόν που εγώ έκανα στην έκθεσή μου είναι ζητάω μια γλωσσα η συμβολα κτλ οχι χρειαζεται πρωτα εκθεση εξολόγηση εξολόγησης εκθεση μου ειναι ζηταω μια μελετη εξολόγηση. προκειμενου να μελετηθούν διάφορα θέματα και μετά να αποφασίσουμε κατά πόσο συμφέρει, κατά πόσο καταναλωτή το θέλει, κατά πόσο είναι εφικτό από τη βιομηχανία να συμμορφωθεί έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ένα πιο απλό σύστημα σήμανσης. Ώστε μόνο οι σημαντικές πληροφορίες να βρίσκονται εκεί και όχι οι πληροφορίες που δεν ενδιαφέρουν τον καταναλωτή, δεν τις χρησιμοποιεί, δεν έχει να τις κάνει. Μερικές φορές οι πολιτικοί θέλουν να προσθέτουν. Ε, λοιπόν, όχι. Τώρα θέλουμε να αφαιρέσουμε. Αλλά ζητάμε από την Επιτροπή, καταρχήν, να μελετήσει κατά πόσο είναι εφικτό να δίνονται πληροφορίες αυτές με έναν άλλο τρόπο. Ζούμε σε μια ψηφιακή κοινωνία. Ίσως οι καταναλωτές που θέλουν να έχουν μια ε, πληροφορία να μπορούν να τη βρουν αλλιώς, σε άλλα επίπεδα. Γι' αυτό και σας το έφερα αυτό εδώ. Να δείτε δηλαδή για ένα μικρό κομμάτι ρούχου πόσες πολλές πληροφορίες, πόσα πολλά πόσες καρτελίτσες έχουμε απάνω για να υπάρχουν οι πληροφορίες που πρέπει να υπάρχουν. Θέλουμε να δώσουμε και χρόνο στην Επιτροπή, δύο χρόνια, γιατί καλή δουλειά χρειάζεται χρόνο για να γίνει. Έπειτα, μιλάμε για την ίνα υφάσματος. Όμως, μερικές φορές υπάρχουν προϊόντα από ζώα που περιλαμβάνονται στα εφάσματα. Ο καταναλωτής δικαιούται να το γνωρίζει αν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αλλά τότε θα πρέπει να προβλέψουμε έναν στάνταρτ ορισμό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως λέμε ότι πρέπει να γίνει και με τα σύμβολα. Τι είναι δέρμα, για παράδειγμα. Εγώ νομίζω ότι το ξέραμε όλοι. Και όμως δεν έχουμε συγκεκριμένο ορισμό για το δέρμα. Δεν ξέρουμε επίσης ποια ευρωπαϊκά προϊόντα ζωικής προέλευσης έχουν δοκιμαστεί και πώς. Δεν υπάρχει και εδώ μια ενιαία προδιαγραφή. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το χρόνο που χρειάζεται για να τα μελετήσει όλα αυτά. Άκουσα από την Επιτροπή πώς θέλουν να το κάνουν, εφόσον τους δώσουμε χρόνο. Ναι, τι λείπει τώρα σε αυτό το σχέδιο έκθεσης. Κάποια θέματα τα αφήνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω εντεταλμένων πράξεων για τις μεθόδους δοκιμής, για τους ορισμούς. Γιατί πρέπει να υπάρχει νομική βεβαιότητα. Αυτό όμως που θέλουμε να πετύχουμε είναι απλοποίηση των ετικετών, της σήμανσης. Μόνο οι αναγκαίες πληροφορίες και όσοι καταναλωτές θέλουν επιπλέον πληροφορίες να έχουν τη δυνατότητα τις πληροφορίες αυτές να τις βρουν αλλού. Όσον αφορά τα οικολογικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, τους κινδύνους για την υγεία κλπ. κλπ. Να, πάλι εδώ σας το δείχνω. Ορίστε, λέει ο κύριος ο οποίος έχει φέρει μαζί του ένα γυναικείο όρουχο. Και κυκλοφορεί στην αίθουσα. Για να... Τα λέω αυτά, λέει ο κύριος για να δείτε πώς ένα τόσο μικρό κομμάτι ρούχου μπορούμε να φορτώσουμε τόσες πολλές ετικέτες. Λοιπόν, στόχος μας είναι να απλοποιήσουμε ώστε και για τη βιομηχανία να είναι τα πράγματα πιο εύκολα, αλλά και να ετοιμάσουμε για το μέλλον την νομοθεσία μας, μην ξεχνάμε ότι ο κόσμος όλο και περισσότερο αγοράζει μέσα από το διαδίκτυο. Χρειάζεται λοιπόν βεβαιότητα και ενημέρωση. Αν όλα αυτά μπορούμε να τα πετύχουμε, τόσο το καλύτερο. Τότε η έκθεσή μου αυτή θα περάσει με ευρύ υποστήριξη. Ελπίζω. Τώρα περιμένω σχόλια από τους συναδέλφους και παρατηρήσεις και από τους κοιόδες εισηγητές βέβαια. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ για τον ενθουσιώδη τρόπο με τον οποίο μας παρουσιάσατε το θέμα σας. Στις 4.30 θα έχουμε εδώ την κυρία Ρέντινγκ. Γι' αυτό και κοιτάω συνέχεια το ρολόι, λέει ο πρόεδρος. Κρέμι, Αλτεμόσα, Ρούλε και Μακάθη είναι στον κατάλογο των ομιλητών. Δεν ξέρω αν και κάποιο άλλος που θέλει το λόγο. Οπότε, δύο λεπτά ας πούμε ο καθένας. Ορίστε εδώ η γραμματεία θα φροντίζει για το ρολόι να δείχνει το χρόνο. Λοιπόν, δύο λεπτά καταρχήν οι παρατηρήσεις σας. Ίσως χρειαστεί περισσότερος χρόνος να παρατείνουμε λίγο την προθεσμία στο κύριο Μάντερς να έχει τη δυνατότητα να συζητήσει το θέμα του περισσότερο με μας. Και η Επιτροπή βέβαια είναι εδώ και θα της δώσουμε το λόγο. Λοιπόν, καταρχήν, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Ήδη ο κύριος Μάντες αναφέρθηκε στις λεπτομέρειες, αλλά εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε έναν από τους στόχους αυτού του ε, κανονισμού, το θέμα της ομοιομορφίας των μεγεθών. Ε, πιστεύουμε ότι το θέμα αυτό των μεγεθών και στην υπόδηση και στην ένδυση είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα ζήτημα το οποίο ε, μας είναι ιδιαίτερος ε, προσφυλές και βεβαίως εμείς δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ε, νέα, νέες απεικονίσεις. Εμείς θέλουμε απλώς να απλουστεύσουμε την διαδικασία και να έχουμε μια ειδική αναφορά ε, εάν πρόκειται για φυσικό υλικό ή για συνθετικό υλικό το οποίο θα ακολουθείται από κάποιο κωδικό. Όσον αφορά τώρα την επισήμανση, συμφωνώ με όσα είπε ο κύριος Μάντερς, δηλαδή είναι απολύτως απαραίτητο να προχωρήσουμε σε απλούστευση ε, και να έχουμε μονάχα αναφορά ε, σε κάποιες επιπλέον πληροφορίες, αλλά με άλλες ε, μεθόδους, όχι δηλαδή με μία επιπλέον ετικέτα πάνω στο ρούχο. Όσον αφορά τώρα το, την αναφορά ε, στην προέλευση, το made in, ε, ναι, εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία τα οποία έχουμε στην διάθεσή μας ε, και οπωσδήποτε δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε καμία αντιπαράθεση πάνω σε αυτό. Όσον αφορά την ιδιαίτερη αναφορά σε ίνες οι οποίες είναι ζωικής προέλευσης, βεβαίως συμφωνώ απολύτως. Ευχαριστούμε πολύ. Η ε, κυρία Μόζα. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Σάντα Να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή που μας έκανε μια πάρα πολύ σωστή αξιολόγηση ε, των πραγμάτων και αναγνωρίσαμε όλοι την, ε, στην παρουσίασή του την συζήτηση ε, που είχαμε κάνει στην Επιτροπή μας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου να διασφαλιστεί η σωστή επισήμανση αυτή άλλωστε ήταν και η ε, πρόταση του παλιού εισηγητού στη διάρκεια της προηγούμενης θητείας. Όσον αφορά ε, τις ετικέτες, βεβαίως θα πρέπει εκεί να γίνεται λόγος ε, στις πρώτες ύλες και γενικότερα συμφωνούμε με όλα αυτά που είπε ο εισηγητής γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε από τι έχει κατασκευαστεί το ρούχο, δηλαδή η πρώτη του ύλη. Ε, βεβαίως ε, κατανοούμε ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε ποιες είναι οι πληροφορίες ε, οι οποίες είναι απαραίτητες για όλους τους καταναλωτές. Τώρα, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όλοι μπορούν να διαβάσουν και να κατανοήσουν τα όσα αναγράφονται στις ετικέτες. Δηλαδή δεν μπορούμε να ε, περιμένουμε ότι ε, κάποιοι καταναλωτές ε, για να καταλάβουν τι αγοράζουν θα πρέπει να πάνε στο διαδίκτυο και να μελετήσουν προσεκτικά. Θα πρέπει όλα να είναι σύντομα, περιεκτικά και κατανοητά. Και βεβαίως να δούμε και πώς μπορούμε να εναρμονίσουμε τα μεγέθη. Και σε αυτό συμφωνούμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ρούλα. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι είναι άσκοπη ενδεχομένω αυτή η μελέτη. Και πραγματικά αυτού του είδους οι εικόνες θα πρέπει να είναι γνωστές, αναγνωρίσιμες και αρκούν. Είμαι κατά, μα πραγματικά κατά, του να μπορεί κανείς να ενημερωθεί περισσότερο μέσω κάποιων άλλων προσβάσεων στο διαδίκτυο ή αλλού. Όταν πραγματικά κανείς έχει πληθώρα πληροφοριών, δεν μπορεί τελικά να έχει σωστή ενημέρωση. Και έχω την εντύπωση ότι ο καθένας από εμά μπορεί να φανταστεί διάφορα παραδείγματα. Ε, είναι πάρα πολύ απλό το τι πληροφορίες χρειάζεται ο κανείς. Πώς πλένεται παραδείγματος χάρη ναι, ένα ρούχο. Ε, η σύνθεση του ρούχου είναι λιγότερο σημαντική για τον καταναλωτή. Βεβαίω, υπάρχουν πολύ σημαντικά πράγματα όπως η απαγόρευση να γίνονται κάποια πειράματα επί των ε, ε, ζώων βεβαίως είτε κάποια ζώα τα οποία δεν θέλουμε να χρησιμοποιούνται αλλά αυτά είναι δεδομένα και πρέπει να απαγορεύονται. Uh, uh, Ευχαριστούμε κυρία Ρούλη και κυρία Μακάρτη. Ευχαριστούμε πρόεδρε. Όπως είπε και ο κύριος Μάντες προηγουμένως, ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι προσπαθούμε να απλουστεύσουμε τις επισημάνσεις, τις ετικέτες ε, και τα αναγραφόμενα σε αυτές. Ε, θα πρέπει να γίνει πιο χρήσιμη η ετικέτα, άρα να περιέχει αυτά τα στοιχεία τα οποία είναι χρήσιμα για, για τον καταναλωτή. Εγώ θα ήθελα να σχολιάσω περισσότερο τα αναγραφόμενα στην τροπολογία 15. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην είμαστε ε, πολύ, να μην πλατιάζουμε με πολλές λεπτομέρειες. Δηλαδή καλύτερα είναι να είμαστε προσεκτικοί έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στην υγεία του καταναλωτή παρά ε, να ε, είμαστε εξαιρετικά ε, αναλυτικοί και βεβαίως θα πρέπει να δούμε και τι λέει και η βιομηχανία, να βοηθήσουμε και τη βιομηχανία σύμφωνα και με τις απαιτήσει των καταναλωτών. Ο κύριος Άριας, ναι, σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Δύο λόγια θέλω να πω, δύο πράγματα. Μιλάμε για την 2020, ε, για τη στρατηγική του 2020. Βρισκόμαστε στην ψηφιακή εποχή και ε, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και να απλουστεύσουμε αλλά να βοηθηθούμε ταυτοχρόνως από τις νέες τεχνολογίες. Ε, στην περίπτωση του ενδύματος ε, το οποίο μας ε, δείχθη εδώ είναι γεγονός ότι οι ετικέτες ήταν πιο μεγάλες από το ίδιο το εσώρουχο εμπροκειμένο. Αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι και στο ίντερνετ μπορούμε να βρούμε κάποιες πληροφορίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον κύριο Ντουράου, εάν ε, θέλει να απαντήσει κυρίως δε στο ερώτημα που έθεσε και ο κύριος Μάντας όσον αφορά την ε, μελέτη αντικτύπου. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος. Πρώτα απ' όλα, ο κανονισμός αυτός αποτελεί και προτίθεται να απλουστεύσει τον υπάρχοντα κανονισμό ε, σχετίζεται ε, μονάχα με, μία, με ένα ε, υποχρεωτικό ζήτημα όσον αφορά συγκεκριμένα την αναγραφή ε, των ινών στην ετικέτα. σε σχέση ε, και με την ε, ε, συνέχιση της διαδικασίας συμφωνούμε να ξεκινήσει συζήτηση μετά την έγκριση της οδηγίας αυτής έτσι ώστε να καλυφθούν όλες οι λεπτομέρειες, οι επιμέρους λεπτομέρειες και βεβαίως να λάβουμε υπόψη την γνώμη των, της κλωστοϊφαντουργίας και όλων των εμπλεκομένων μερών. Εκεί λοιπόν μπορεί να υπάρξει η μελέτη αντικτύπου έτσι ώστε να δούμε εάν μπορούν να αναλυφθούν κάποιες ε, πρωτοβουλίες εάν αυτό καταδειχθεί μετά ε, τις ε, συζητήσεις. Όμως καταρχάς η αναφορά στα, στα ζωικής, στη ζωική πρόέλευση ή πιστεύω ότι θα πρέπει πρώτα να γίνει ύλης πιστεύω ότι θα πρέπει πρώτα να γίνει η μελέτη και μετά να παρουσιάσουμε όλες τις επεξηγήσεις αν δηλαδή θα πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα πιο πέρα ή αν ε, θα πρέπει να σταματήσουμε εδώ. Εάν κατάλαβα καλά, λέει ο Πρόεδρος, αυτό που είπατε, θέλετε να συνεχίσουμε με βάση αυτήν την πρόταση και οποιαδήποτε περαιτέρω εξέταση να γίνει μετά. Δηλαδή να μην, ε, να μην κάποια πρωτοβουλία τώρα. Αυτό για να είμαστε όλοι σαφείς. Ναι, ναι, ε, κύριε Πρόεδρε. Αυτή είναι η άποψή μας. Θεωρούμε δηλαδή ότι το, καλό, το καλύτερο θα ήταν να ε, γίνει μία ε, διόρθωση όσον αφορά τις απαιτήσεις αναγραφής των ετικετών αλλά ότι δεν υπάρχει λόγος να αλλάξουμε εκβάθρον όλο το σύστημα. Ε, πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι έχουμε εκπρόσωπο και της Προεδρίας. Δεν ξέρω εάν ε, θέλει να πάρει το λόγο. Ναι, παρακαλώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, ήθελα απλά να σας πω ότι στο Συμβούλιο εμείς έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει την επεξεργασία του κειμένου και ε, ε, παραμένουν κάποιες ε, λεπτομέρειες όπου το Κοινοβούλιο έχει επιφύλαξη σκέψης και πέρα από αυτό νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Βεβαίως θα μελετήσουμε και τα αποτελέσματα της μελέτης και εν πάση περιπτώσει εμείς θα θέλαμε η συζήτηση σχετικά με την αύξηση των στοιχείων ε, που πρέπει να αναγράφονται στις ετικέτες, κυρίως όσον αφορά την σύνθεση των ινών, ε, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης αντικτύπου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατά τα λοιπά, θα θέλαμε το προτινόμενο κείμενο να τεθεί σε ισχύ όσο γίνεται πιο ε, πολύ. Βεβαίως ε, είμαστε διατεθειμένοι να εργαστούμε στενά με τον εισηγητή και τον σκιώδη εισηγητή έτσι ώστε να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα ε, όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ο εισηγητής κ. Μέντες μήπως θέλει σύντομα να ολοκληρώσει να κάνει μια τελευταία δηλαδή ε, παρουσίαση. Ο κύριος Μάντερς, ευχαριστώ πολύ. Άκουσα όλους τους παρεμβαίνοντες και νομίζω ότι όλοι είναι πεπισμένοι πλέον ότι θέλουμε απλούστευση ε, των ετηγετών, Θέλουμε μεγαλύτερο βαθμό ε, ε, μεγαλύτερο βαθμό πιστοποίησης και ομοιομορφίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θέλουμε δηλαδή τα πρότυπα να είναι όσο γίνεται πιο εναρμονισμένα. Και επομένως μέσω της μελέτης μπορούμε να καταλήξουμε στο που πώς μπορούμε να ε, έχουμε μια σήμανση η οποία θα δίνει ακριβώς τα στοιχεία που χρειάζονται. Ε, τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Ε, νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, Ξέρετε ότι υπάρχει χρονοδιάγραμμα για τις τροπολογίες. Ναι, έχω προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 19 Μαρτίου, δηλαδή το τέλος της εβδομάδας. 7 Απριλίου τελική συζήτηση, 8 Απριλίου τελική ψηφοφορία. Εάν όλοι συμφωνούν, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε με το χρονοδιάγραμμα αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, λοιπόν, 19 Μαρτίου στις 2 το μεσημέρι προθεσμία υποβολής ε, τροπολογιών, συζήτηση 7 Απριλίου, ψηφοφορία 8 Απριλίου. Ωραία λοιπόν, μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο και πρέπει να πω ότι με μεγάλη χαρά έχουμε, ε, μπορούμε να υποδεχθούμε την δεύτερη αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπεύθυνοι για νομικές υποθέσεις αλλά και ένα σωρό άλλα ε, ζητήματα τα οποία ιδιαιτέρως ε, μας είναι προσφυλή και μας απασχολούν. Ε, η Επίτροπο κυρία Vivian Ρέντινγκ, η οποία βεβαίως είναι παλιά γνώριμη της Επιτροπής Ξέρουμε ότι στην προηγούμενη θητεία της Επιτροπής ήταν μια πολύ επιτυχημένη επίτροπος για θέματα πληροφορικής και τα λοιπά, για την ε, κοινωνία της πληροφορίας και βεβαίως πριν από αυτό ήταν εδώ μαζί μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι, πρέπει να σας πω επίσης ότι είμαστε μαζί χθε στην ε, Μαδρίτη. Ε, ξέρω ότι έχετε κάποια καινούργια στοιχεία να μας πείτε. Με μεγάλη χαρά λοιπόν θα σας δώσουμε το λόγο και μετά θα ακούσουμε τις απόψεις των συναδέλφων. Ξεκινήσουμε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 αναμίχθηκα ιδιαιτέρως και ενδιαφέρθηκα ιδιαιτέρως για θέματα προστασίας του ε, καταναλωτού και βεβαίως ε, από πολύ κοντά είδα κυρίως το θέμα των τελειπικοινωνιών έτσι ώστε ε, αυτές να γίνουν πιο φιλικές προς τον καταναλωτή, πιο εύκολα προσβάσιμες κλπ. Έχουμε δουλέψει πολλές φορές ε, σε σύμπνοια με το Κοινοβούλιο και για την οδηγία των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε ε, με πολύ αποφασιστικά βήματα όσον αφορά ε, την νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών, ξεπερνώντας τα όποια προβλήματα ή όποιες αντιδράσεις. Ξέρω ότι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλετε να γνωρίζετε όλες τις επιπτώσεις που θα έχει το κείμενο αυτό ε, στους καταναλωτές και οι συζητήσεις σας προς αυτήν την κατεύθυνση οδεύουν. Ο διάλογος λοιπόν είναι εξαιρετικά σημαντικός και θα πρέπει να ενισχυθεί. Πιστεύω ότι κυρίως σε καιρούς κρίσης πρέπει να ενδυναμώσουμε την αίσθηση του καταναλωτή ότι όταν ε, ε, ψωνίζουν ακόμα και διασυνοριακά ότι προστατεύονται τα δικαιώματά τους όταν κάνουν τις αγορές τους δηλαδή να έχουν μια αίσθηση ασφάλειας και προστασίας ε, των καταναλωτών. Γι' αυτό λοιπόν έχετε το κείμενο αυτό μπροστά σας. Ένα κείμενο το οποίο είναι ηθελημένα φιλόδοξο γιατί ζητάει να προχωρήσουν ε, όλες οι διαδικασίες έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια πραγματικά ενιαία αγορά όσον αφορά την προστασία των ε, δικαιωμάτων των ε, καταναλωτών. Θέλουμε να λειτουργεί καλά η αγορά, αλλά θέλουμε να έχουν και αίσθηση δικαίου οι καταναλωτές και γνωρίζετε ότι όταν ας πούμε, μιλάμε ε, για το διαδίκτυο, εκεί η εσωτερική αγορά σταματάει. Σε μια έρευνα που κάναμε, κατεδείχθη ότι 61% και τονίζω 61% των διασυνοριακών ε, online ε, συναλλαγών δεν ολοκληρώνεται γιατί δεν υπάρχει υποστήριξη Ξέρετε ότι εμείς στο Λουξεμβούργο είμαστε ε, μια μικρή χώρα ε, και επομένως ε, και για να κουνήσουμε που λέει ο λόγος το μικρό μας δαχτυλάκι θα, βρεθούμε, θα πρέπει να βρεθούμε σε μια άλλη χώρα, θα πρέπει να περάσουμε τα σύνορα. Πρέπει να πω επίσης ότι μονάχα 12% των χρηστών του δικτύου, του διαδικτύου στην Ευρωπαϊκή Ένωση αισθάνονται ασφαλής και εδώ δεν έχει να κάνει μονάχα με το διασυνοριακό εμπόριο, ακόμα και για το εμπόριο στην ε, εσωτερική τους αγορά. 12% συνολικά των χρηστών του διαδικτύου αισθάνονται ασφάλεια και είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν το ε, διαδίκτυο ε, το διαδίκτυο για τις αγορές τους αλλά φοβούνται ε, και ξέρετε αυτή η έλλειψη ολοκλήρωσης της εσωτερικής online αγοράς κοστίζει εκατομμύρια ευρώ χάνουμε πάρα πολλά και νομίζω ότι είναι κρίμα. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να χάσουμε αυτήν την εμπορική ε, ευκαιρία. Επομένως, χρειαζόμαστε εναρμόνιση. Ξέρουμε ότι εάν έχουμε ήδη ομοιόμορφα δικαιώματα ε, καταναλωτών, οπωσδήποτε θα αποτελεί ένα ε, καλό πρώτο βήμα και βεβαίως ε, θα δυναμώσει την εμπιστοσύνη των πολιτών είτε στην εσωτερική τους αγορά, είτε στις διασυνοριακές τους ε, συναλλαγές. Ε, θα μπορούσαμε ενδεχομένως να κάνουμε και κάποια ε, πανευρωπαϊκή εκστρατεία πληροφόρησης έτσι ώστε να πάψει ο κατακαιρματισμός της αγοράς αυτής και ο κατακαιρματισμός των δικαιωμάτων. Το σημαντικό είναι να αισθάνονται οι πολίτες εμπιστοσύνη έτσι ώστε να αγοράζουν και στη δικιά τους αγορά αλλά και στο εξωτερικό η οδηγία δικαιωμάτων των καταναλωτών είναι πάρα πολύ σημαντική και ο υψηλός βαθμός προστασίας των καταναλωτών θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στο κείμενο. Βρίσκεται εδώ όμως το κείμενο. Όπως και να σα το πω η απάντηση είναι όχι. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω ε, τα, τον προβληματισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και αυτών των κρατών μελών. Καταλαβαίνω βεβαίως ότι η πλήρης εναρμόνιση θα σήμαινε για κάποιες ε, χώρες μέλη ότι θα πρέπει να προσαρμόσουν προς τα κάτω την προστασία των καταναλωτών του σε επίπεδο δηλαδή χαμηλότερο από αυτό που έχουν αυτή τη στιγμή και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το εξηγήσει κανείς. Πώς είναι δυνατόν ε, να εξηγήσει κανείς σε κάποιον πολίτη α πούμε ότι ναι ξέρετε κάνουμε μια οδηγία για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών αλλά αυτό θα σημαίνει ότι τα δικιά σα δικαιώματα θα είναι λιγότερα πλέον από ό,τι είχατε μέχρι τώρα. Είναι, είναι πολύ λεπτό το ζήτημα. Το πιο εύκολο βεβαίως, η πιο εύκολη λύση θα ήταν ότι ανεβάζουμε το επίπεδο όλων. Δεν είμαι όμως σίγουρη ότι όλα τα κράτη-μέλη θα θεωρούσαν ότι αυτό είναι προφανές και εύκολο. Είναι πάντως σαφές ότι δεν υπάρχει ε, σωστό επίπεδο προστασίας ε, σε όλες τις ε, χώρες. Συμφωνώ με αυτό και συμφωνώ ε, να υπάρξουν περαιτέρω συζητήσει με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. και διάβασα το έγγραφο εργασία του εισηγητού σα Ανδρέα Σουάμπ ε, που πραγματικά εξηγεί ότι το, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθεί με κάθε δυνατό και δημιουργικό τρόπο να βρει μια ισορροπημένη ε, λύση και μάλιστα η πρόταση εναρμόνισης της Κομισιόν του 2008 ε, έχει θέσει τους σωστούς στόχους έτσι ώστε να λύσουμε τα προβλήματα τα οποία σχετίζονται με την ε, εσωτερική ε, αγορά αλλά βεβαίως θα πρέπει να βρούμε και κάποιες πιο πρακτικές λύσεις. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε και το ενδεχόμενο της πιο στοχευμένης εναρμόνισης. Μία πιθανότητα θα ήταν να προχωρήσουμε με πλήρη εναρμόνιση όσον αφορά τις ε, συμβάσεις εξ ε, και να συγκεκριμενοποιήσουμε το περιεχόμενο αναπερίπτωση. Όσον αφορά τώρα ε, τις συναλλαγές online, ενδεχομένως θα μπορούσαμε σε μια δεύτερη φάση να ζητήσουμε ε, μεγαλύτερη εναρμόνιση με τα offline, με τις offline συναλλαγές, αλλά αυτό μπορεί να γίνει λίγο αργότερα. Αφήστε με να σας παρουσιάσω τα κύρια σημεία για να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Υπάρχουν πέντε κύριοι τομείς που δεν έχουν όλη την ίδια δυσκολία βεβαίως. Πρώτος τομέας. Ορισμοί. Ξέρω ότι εργαστήκατε σκληρά για το θέμα του ορισμού, το ίδιο και το Συμβούλιο, έτσι ώστε να υπάρξουν ε, συνεκτικοί κανόνες και πραγματικά πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε με αισιοδοξία βλέπω αυτό το σημείο και να οδηγηθούμε σε εναρμονισμένους ορισμούς αυτό είναι, αν θέλετε, το πιο εύκολο κομμάτι όλου αυτού του εγχειρήματο. Ξέρω ότι κάποιοι είναι υπέρ της αμοιβαίας αναγνώρισης. Εγώ δεν είμαι σίγουρη. Καθότι η αμοιβαία αναγνώριση μπορεί να είναι λύση για τις επιχειρήσεις, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε νομική αβεβαιότητα τους καταναλωτές. Και εκεί κινδυνεύουμε να οδηγηθούμε σε έναν ε, νομικό κατακαιρματισμό, ε, κάτι που θα πρέπει να αποφύγουμε. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι εδώ πραγματικά δεν είμαι σίγουρη. Δεύτερο, όσον αφορά την προσυμβατική ενημέρωση, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν χώρες που έχουν πολύ συγκεκριμένους ε, κανόνες για θέματα υγείας, κάτι που θα πληγεί σοβαρά από την πρόταση αυτή. Πρέπει λοιπόν να είμαστε εξαιρετικά ρεαλιστές, πραγματιστές και να επικεντρωθούμε σε όλους αυτούς τους τομείς που έχουν πολύ σημαντική διάσταση όσον αφορά την εσωτερική αγορά. Επίσης, όσον αφορά τις άμεσες συμβάσεις. θα πρέπει συμβάσεις που συνάπτονται από τα ίδια τα φυσικά πρόσωπα. Πρέπει λοιπόν εδώ να εναρμονίσουμε σαφώς όλους αυτούς τους κανόνες έτσι ώστε οι άμεσες συναλλαγές αλλά και οι εξαποστάσεως συναλλαγές να διεκπεραιώνονται βάσει των κανόνων των χωρών αλλά και σε διασυνοριακό επίπεδο και ξέρουμε σήμερα ότι υπάρχουν παραδείγματο χάρη οι 40 ημέρες η προθεσμία που σαφώς θα πρέπει να διατηρηθεί για να κρατηθεί αυτή, αυτό το επίπεδο νομικής ε, ασφάλειας. Και εδώ θα πρέπει να κάνουμε μία διάκριση. όσον αφορά την ε, παραλλαγή των προϊόντων, την παραλαβή των προϊόντων, όσον αφορά την αποστολή, όσον αφορά τους κανόνες, ε, διαφέρουν πάρα πολύ από τη μια χώρα στην άλλη. Παραδείγματο χάρη, για περίπτωση απώλεια ενό προϊόντος που αποστέλλεται στον καταναλωτή, είτε για βλάβε, θωρά, ο υπεύθυνο δεν είναι ο ίδιος ανάλογα με το σε ποια χώρα βρισκόμαστε. Παραδείγματο χάρη στην Ιταλία προστατεύεται πολύ περισσότερο ο καταναλωτή. Υπάρχουν λοιπόν εδώ πολλές και διαφορετικές προσεγγίσεις και είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί μέση οδό όσον αφορά τις αποζημιώσεις, όσον αφορά τις νομικές εγγύησεις. Επίσης η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική καθότι η σχέση μεταξύ του συμβατικού δικαίου και των αποζημιώσεων που προβλέπονται για τον καταναλωτή είναι τελείως διαφορετικές. Παραδείγματο χάρη, στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί κάποιο να στείλει πίσω ένα προϊόν. Στην Γαλλία υπάρχουν εγγύησει για κάποια ελαττώματα που δεν φαίνονται καταρχήν, αλλά ανακαλύπτει ο καταναλωτής καθυστερημένα. Πλήρης εναρμόνιση λοιπόν είναι κάτι που δεν θεωρώ ότι μπορεί να γίνει εύκολα, δεν είναι ρεαλιστική. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ παραδείγματος χάρη των συμβάσεων αυτών που εμπίπτουν στην ενή αγορά και των συμβάσεων αυτών που ονομάζουμε άμεσες συμβάσεις. Και πιστεύω πραγματικά ότι εδώ θα πρέπει να γίνουν διαπραγματεύσεις. Όσον αφορά τους αθέμητους όρους που μπορεί να περιέχει μία σύμβαση. Εάν θεωρήσουμε ότι πρέπει να υπάρξει μία ρήτρα όσον αφορά ε, τον αθέμητο, τους αθέμητους όρους, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει τα δικαστήρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουν την εξέταση για το αν υπάρχουν ή όχι τέτοιοι ε, όροι και θα πρέπει να τηρηθούν εδώ τα ίδια κριτήρια για να γίνει η αξιολόγηση αυτών των συμβάσεων και των διατάξεων. Η αξιολόγηση λοιπόν θα πρέπει να γίνει βάσει των ίδιων κριτηρίων. Άρα πηγαίνουμε προς μια πλήρη εναρμόνιση. Το ερώτημα λοιπόν είναι, και αυτό είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον, είναι να υπάρξει ένας κατάλογος των αθέμητων ή παράνομων όρων για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο δεν μπορεί να υιοθετηθεί σε εθνικό επίπεδο. Και εδώ υπάρχει μία εναλλακτική λύση. Να υπάρχει δηλαδή ένας τέτοιος κατάλογος μόνο για τις εξαποστάσεως εμπορικές συναλλαγές και όχι για την άμεσες εμπορικές συναλλαγές και συμβάσεις. Πρόεδρε, πρόκειται για μια πρόταση προφορική από μέρος της Επιτροπής, την γραπτή την έχετε, αλλά πρόκειται για μια πρόταση που έχει σαν σκοπό να βγούμε από το αδιέξοδο. Και όλοι οι νομοθέτες, οι νομοθετικές αρχές να συνεργαστούν έτσι ώστε να βρεθεί μια λύση που να ικανοποιεί και τον καταναλωτή και τις επιχειρήσεις. Γιατί πιστεύω ότι δεν είναι αντικρουόμενα τα συμφέροντα των μεν και των δε και ότι στις τελικές μας διαπραγματεύσεις θα πρέπει να υποβληθεί ένα καλό κείμενο το οποίο να είναι προς συμφέρον και των δύο αυτών ομάδων. Δείχνω λοιπόν με αυτή την πρόταση ένα πνεύμα ανοιχτό έτσι ώστε να βελτιωθεί το κείμενο και να εργαστούμε περαιτέρω. Ευχαριστούμε πολύ για όλες αυτές τις λεπτομέρειες που μας δώσατε. Μας μιλήσατε για το μέλλον. Πού πρέπει να κατευθυνθούμε. Για να δούμε οι συνάδελφοι τι έχουν να πούν για όλα αυτά. Προτείνω, γιατί είσαστε εδώ τουλάχιστον μέχρι τις 5.30, έτσι δεν είναι. Έχουμε χρόνο, νομίζω, για να έχουμε μια καλή συζήτηση. Οπότε, κάθε τρεις ερωτήσεις θα απαντάει μετά η Επίτροπος. Έχω πέντε σκιώδεις, ΣΦΑΠ, ΚΕΠΑΡΤ, Ρόσφορτ, Τούρνεν και Τρενταφυλλίδης. Και μετά Σαλτεμόσα, Μπουζόη, Κορέντε Κάπο, Στέιλερ, Βέρτιο και η κυρία Ράπτη. Και την κυρία Ρούλε. Άλλος κανείς και ο κύριος Έλιας. Λίγο πολύ όλοι. Καλώς τρεις ερωτήσεις μαζί και παρακαλώ να είσαστε ακριβείς όσον αφορά το θέμα της ερώτησής σας για να μπορέσει να απαντήσει καλά και η Επίτροπος και έτσι να έχουμε έναν ωραίο διάλογο. Σβάπ, Κέπαρτ και Ρόσφορτ είναι οι πρώτοι τρεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ την Αντιπρόεδρο εξ ονόματος του ΕΛΚ. Θα ήθελα να σας πω ότι πραγματικά εκτιμάμε ιδιαίτερα το ότι ταχύτατα αντιδράσατε και κάνετε αυτήν την πρόταση Πρόκειται για ένα θέμα που φυσικά και ο προηγούμενος Επίτροπος είχε επεξεργαστεί. Είναι ένα θέμα που αφορά άμεσα τα συμφέροντα των καταναλωτών. Από την άλλη μεριά βεβαίως η εσωτερική αγορά, η νέα αγορά και οι ευκαιρίες και δυνατότητες που προσφέρει για τους καταναλωτές στην Ευρώπη. Ξέρω ότι εχθές ε, στη Μαδρίτη αναφερθήκατε στο θέμα και μιλήσατε για τις βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν χωρίς βεβαίως την ίδια ώρα να δημιουργήσουμε εμπόδια και προσκόμματα για τις επιχειρήσεις. Και εγώ σαν εισηγητής δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να είμαι αντίθετος με την ιδέα ότι τίποτα δεν πρέπει να εμποδίσει τα συμφέροντα ε, και την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών. Λαμβάνεται λοιπόν πάρα πολύ σοβαρά εδώ αυτές τις αρμοδιότητες όπως και εμείς και πιστεύω ότι θα πρέπει από κοινού να βρεθεί μία πρόταση, ένα κείμενο που να είναι αποδεκτό και από το Συμβούλιο. Καταρχήν λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να συνεισφέρουν, να συμμετέχουν. Στο κεφάλαιο 5 υπάρχουν διάφορες δυνατότητες. Ξέρω ότι και με τους συνεργάτες σας έχουμε συζητήσει τα θέματα αυτά, αλλά αυτό που είναι ε, πολύ ενδιαφέρον να δούμε εδώ ότι πολλοί ανησυχούν ε, στην Ευρώπη σε όλους τους τομείς όσον αφορά την ε, ενοποίηση και επίτηδες θα χρησιμοποιώ άλλο όρο την ενιοποίηση η οποία μπορεί να προσθέσει ακαμψία και αυτό το ακούμε και από μέρους των καταναλωτών αλλά και από μέρους των επιχειρήσεων. Δεν πρέπει επουδενή λόγο εδώ να οδηγηθούμε σε νέα αρνητικά, αν θέλετε, σχήματα τα οποία θα είναι αρνητικά και για τους καταναλωτές αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι πολλοί εμπειρογνώμονες της Επιτροπής έχουν εκφράσει τέτοιες απόψεις. Η ερώτησή μου λοιπόν ε, βεβαίως έχει άμεση σχέση με αυτό. Το δεύτερο σημείο που εσείς αναφέρατε είναι ο διαχωρισμός μεταξύ των διαφόρων εμπορικών συναλλαγών offline, online και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θέλετε να συνεχιστεί η επεξεργασία του θέματος αυτό σε διμέρες επίπεδο. Ξέρω ότι στην Μαδρίτη είπατε ότι πολλοί καταναλωτές βλέπουν κινδύνους σε αυτές τις εμπορικές συναλλαγές, ιδιαίτερα όταν παραδείγματο χάρη γίνονται αγορές online, όταν κάποιος βρίσκεται απέναντι σε έναν πολιτή, όταν γίνεται δηλαδή μια άμεση εμπορική συναλλαγή, υπάρχουν πολλά σήματα, όπως ε, ακόμα και η αντίδραση, η σωματική, ο τρόπος που κάποιος δείχνει την αμηχανία του ή όχι, που μπορούν να αυξήσουν την εμπιστοσύνη αυτού ο οποίος καλείται να αγοράσει ένα προϊόν. Θα ήθελα λοιπόν πραγματικά να φτάσουμε σε ένα αποδεκτό αποτέλεσμα, κάτι το οποίο να καθησυχάζει και να προστατεύει τα συμφέροντα των Ευρωπαίων καταναλωτών. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σουάπη, κυρία Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ρέντινγκ για την σημερινή σας παρουσίαση και τις απαντήσεις που προτίθεται να δώσετε στις ερωτήσεις μας. Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό θέμα και αυτό που θα ήθελα εγώ να σας αναφέρω είναι ότι πραγματικά είμαι για την πλήρη εναρμόνιση. Αυτή ήταν η πρώτη μου αντίδραση και κατόπιν βεβαίως ήρθαμε σε μια νέα θέση, υιοθετήσαμε μια νέα θέση όσον αφορά την εναρμόνιση και την προστασία κάποιων δικαιωμάτων. Ξέρω, παραδείγματο χάρη, ενώ και αυτό αφορά το Λουξεμβούργο, ότι οι καταναλωτές δεν θέλουν να υποχωρήσουν σε ένα τμήμα των δικαιωμάτων τους, στην προστασία κάποιων από τα δικαιώματά τους και εσείς βεβαίως υποστηρίξατε αυτή τη θέση. Σε αυτό το σχέδιο το οποίο μας έχει υποβάλει εδώ η Επιτροπή βλέπουμε ότι τα δικαιώματα των καταναλωτών υποβαθμίζονται και αυτό επουδενή λόγο δεν θέλουμε εμείς να το δεχτούμε. Το ερώτημα λοιπόν είναι αυτό το σχέδιο νομοθετικού κειμένου για να εγκριθεί από όλους θα πρέπει να τροποποιηθεί πάρα πολύ και σε πάρα πολλά σημεία. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξή. Είστε διατηρημένοι να αποσύρετε το κείμενο αυτό έτσι ώστε βάσει ενός πιο λογικού κειμένου, μιας πιο λογικής πρότασης να εργαστούμε γιατί πραγματικά το παρόν κείμενο είναι πάρα πολύ δύσκολο να ε, το επεξεργαστούμε και να το αλλάξουμε. Η απάντησή σας όμως είναι όχι από ό,τι κατάλαβα και πραγματικά θα αναγκαστούμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτό το κείμενο το οποίο δεν είναι τόσο καλό. Άρθρο 4, και αυτό είναι το τρίτο σημείο που θα ήθελα να δείξω, η πλήρης εναρμόνιση. Τα δικαιώματα τα οποία σήμερα υπάρχουν σε κάποια κράτη-μέλη και τα οποία είναι ισχυρότερα από αυτά που προτείνει το κείμενο αυτό. Δηλαδή μιλάμε για μια υποβάθμιση και σε αυτό εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να υποχωρήσουμε. Αυτή η υποβάθμιση των δικαιωμάτων είναι κάτι που πραγματικά δεν θέλουμε να το δεχτούμε. Θέλουμε να συνεχίσουμε να προστατεύουμε στον ύψιστο βαθμό τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Και εμείς σαν social δημοκράτες θα σας ακολουθήσουμε και θέλουμε να προχωρήσουμε σε ένα λογικό και αποδεκτό κείμενο. Ευχαριστούμε για αυτά τα πολύ ξεκάθαρα που μας είπατε. Ο κύριος Ροσφόρ έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ σήμερα που η Επιτροπή μας μεταφέρει μέσω ημών ένα μήνυμα δημιουργικότητας. Βλέπετε εδώ και πολύ καιρό, εδώ και πολλούς μήνες είμαστε σε δύσκολη θέση και εσείς σήμερα μας φέρνετε κάποια νέα στοιχεία, κάποιες νέες προτάσεις που πιστεύω ότι αποτελούν ένα μικρό δείγμα αλλαγή στον προσανατολισμό του τι εννοούμε με το ανώτατη αναρμόνιση Νομίζω ότι αυτά που προτείνετε είναι ενδιαφέροντα πράγματι. Συνήθως μιλάμε για την εξαποστάσεως αγορά που γίνεται όχι μόνο μέσω διαδικτύου και μέσω τηλεφώνου μερικές φορές ή με το ταχυδρομείο. Αυτή η πώληση και αγορά δεν είναι της ίδιας φύσης όπως εκείνη που γίνεται τέτα τέτ. Οπότε, αν αποσύρουμε πολλά από αυτά που έχουν να κάνουν με την άμεση πώληση όσον αφορά την ανώτατη προστασία. Αυτό δεν οδηγεί τον ε, καταναλωτή σε περισσότερη αδυναμία. Από ό,τι φαίνεται είναι περισσότερο σε αδυναμία, είναι πιο ευάλωτο σε μια απευθείας συναλλαγή παρά σε συναλλαγή εξ αυτή η συναλλαγή λοιπόν εξ αποστάσεως είναι μια εξέλιξη σίγουρη. Εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρος αν τα νούμερα που ακούμε είναι πραγματικά. Πάντως όσον αφορά την άμεση αγορά και πώληση υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τυποποιήσει τις πωλήσει τους σε διάφορες χώρες μέλη. Παρόλο που μέχρι τώρα ξέραμε μια τέτοια τυποποίηση μόνο στις εξαποστάσεις. Φανταστείτε έναν Πορτογάλο να αγοράζει στη χώρα του ένα Ιρλανδό στη δικιά του με τον ίδιο τρόπο. Γίνεται όταν έχουμε μέσω διαδικτύου αγοροπολισία συναλλαγή, τότε ναι. Αυτή η τυποποίηση της συναλλαγής είναι λογική. Υπάρχουν ένα σωρό θέματα πάντως, πολλά από τα οποία εξηγούνται πάρα πολύ καλά στο σχέδιο έκθεσης του κυρίου Σφάμπ. Το γνωρίζετε κι εσείς το έγγραφο αυτό. Εννοείται ότι μένουν πολλά να διακανονιστούν ακόμα. Παραμένει πολλή δουλειά να γίνει. Ακόμα κι αν θεωρείτε ότι όσον αφορά την ανώτατη εναρμόνιση, εσείς επικεντρωνόσαστε στην εξαποστάσεως αγοροπολισία. Εγώ πιστεύω ότι όλη η δουλειά μένει να γίνει ακόμα. Γιατί υπάρχουν ιδιαιτερότητε σε διάφορα είδη πώληση προϊόντων. όπω επίση όσον αφορά τη διάρθρωση, το δίκαιο δηλαδή το οποίο εφαρμόζεται στα πλαίσια αυτή τη οδηγία ισχύει και στι συμβάσει, Εγώ δεν ξέρω αν αυτή τη διάκριση που εσείς προτείνετε πρέπει εμείς να τη δούμε σαν πανάκια. Εγώ νομίζω ότι τα προβλήματα παραμένουν. Και για παράδειγμα, Κάτι που μου έκανε εντύπωση στην έκθεση ΣΦΑΠ είναι ότι σε κάθε κεφάλαιο ζητάει επιπλέον μελέτες αξιολόγησης. Αυτό τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας. Είμαι λοιπόν πεπισμένος γι' αυτό. Πάντως εκτίμησα πολύ ε, το γεγονός ότι χρησιμοποίησατε τη λέξη πραγματισμός, ρεαλισμός, γιατί όντως περί αυτού πρόκειται. εξαρτάται από το πώς θα κρατήσουμε τα γέμια. Εσωτερική αγορά για τις επιχειρήσεις και εμπιστοσύνη για τον καταναλωτή. Αυτά τα δύο είναι που πρέπει να χειριστούμε καλά για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Θα ήταν λοιπόν ενδιαφέρον η ισορροπία να υπάρχει ξεκάθαρα και να το βλέπει ο καταναλωτής να είναι αυθεντική η προστασία του καταναλωτή. Στην αρχή το είπατε αυτό. Εγώ θα ήθελα να φαίνεται και παντού ότι είναι έτσι. Ευχαριστώ. Ωραία. Η Επίτροπος να απαντήσει στις τρεις πρώτες ερωτήσεις τώρα. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που είναι σημαντικό γενικά μιλώντας είναι η Επιτροπή να μην επιμείνει κατά λέξη στο αρχικό κείμενο. Τώρα, το να πούμε ότι θα ξεκινήσουμε από το μηδέν, ε, νομίζω ότι είναι υπερβολικό. Κυρίως γιατί σε επίπεδο Συμβουλίου και σε επίπεδο Κοινοβουλίου έχει ήδη γίνει πολλή δουλειά. Αυτό που ήθελα να πω με τα διάφορα άρθρα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ελαστική συνοδεύει τη δουλειά που γίνεται τόσο στο Συμβούλιο όσο και στο Κοινοβούλιο με ανοιχτό πνεύμα. Δεν θα αντιτεθούμε σε προτάσεις οι οποίες αντιβαίνουν στο βασικό κείμενο. Όμως, για να μην επαναλάβουμε ξανά μια δουλειά που στο κάτω-κάτω δεν είναι εύκολη, γιατί το βασικό κείμενο το έχουμε από το 2008 είμαστε 2010. Ε, ναι. Οπότε κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη στον νομοθέτη. Και μετά, με τα ταπεινοφροσύνη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πριν τη δεύτερη ανάγνωση, θα προτείνει ένα νέο κείμενο. Όμως, Ειλικρινά, θα ήθελα και τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλοι οι εμπλεκόμενοι, οι stakeholders, να έρθουν με προτάσεις κειμένου. Εισαγωγικά είπα ότι δεν μπορώ να φανταστώ να έχουμε ένα κείμενο προστασίας των καταναλωτών που να μην προστατεύει τελικά τους καταναλωτές. Και γι' αυτό τι χρειάζεται. Πρέπει κάθε φορά να διαγραφεί η πλήρης αναρμόνιση. Δεν είναι βέβαιο. Γιατί εκεί όπου μας εξυπηρετεί μπορούμε να την κρατήσουμε. Εκεί όπου προστατεύει τον καταναλωτή πρέπει να την κρατήσουμε. Εκεί που αντίθετα πλήττει το καταναλωτή, όχι. Για μένα δεν είναι ιδεολογικό το ζήτημα. Είναι ρεαλισμός να προσπαθήσουμε να βρούμε τις καλύτερες λύσεις. Εννοείται ότι το ιδεώδες, το ιδανικό θα ήταν να έχουμε μια πλήρη εναρμόνιση στο ανώτατο. Έτσι. Δεν νομίζω όμως ότι θα συμφωνούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ενώ πρέπει να υπάρξει συμφωνία Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Αυτό λοιπόν που θα μπορούσα να κάνω σε αυτό το στάδιο είναι να βάλω και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στη σωστή κατεύθυνση και από εκεί και πέρα αν το ζητήσουν οι νομοθέτες, να προτείνουμε για δεύτερη ανάγνωση μια νέα πρόταση. Τώρα για τις μελέτες ε, αντικτύπου. Ο κύριος Ροσφόρ είπε ότι ο κύριος Βαπ θέλει περισσότερες μελέτες αντικτύπου. Ναι. Ωραία. Οπότε, αν είναι αναγκαίο, ναι. Αλλά εγώ δεν θέλω να κάνω μελέτες αντικτύπου για το τίποτα, χωρίς λόγο. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Έπειτα είναι και χρονοβόρο. Εάν ήταν αναγκαίο, δεν θα έλεγα όχι. Πάντως νομίζω ότι γνωρίζουμε όλοι περί τίνος πρόκειται. Και αν δεν κάνουμε επαναστατικές προτάσεις, είναι προτιμότερο να αποφεύγουμε τέτοιες μελέτες αντικτύπου. Εγώ είμαι υπέρ συγκεκριμένων προτάσεων που θα δοκιμαστούν. Πρώτα απ' όλα για να δούμε ποια είναι η γνώμη των άμεσα ενδιαφερομένων. Σε μια τέτοια οδηγία, τέτοιου είδου πρέπει να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στα συμφέροντα των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, των εμπόρων. Ισορροπία χρειάζεται. Ακόμα και αν πρόκειται για ένα κείμενο το οποίο αναφέρεται στην προστασία των καταναλωτών. Αλλά η προστασία του κλάδου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι επίσης κάτι το αναγκαίο. Έπειτα, πρέπει ο καταναλωτής να έχει εμπιστοσύνη. Είναι τετραγωνισμός του κύκλου. Θα τα καταφέρουμε όμως, πιστεύω. Οπότε ξεκάθαρα θέλω να σας πω ότι πρέπει τα διάφορα προβλήματα να τα δούμε ένα-ένα. Και υπάρχει και κάτι το οποίο δεν το έχω καταλάβει καλά. Κύριε Σβάμπ. Εφόσον έχουμε μια οδηγία, θα έχουμε πληροφορίες από τους καταναλωτές, από τον κλάδο επίσης και από εκεί και πέρα πώς μπορούμε να αλλάξουμε την οδηγία βάσει αυτών των πληροφοριών. Για μένα είναι λεπτό το ζήτημα. Άπαξ και έχει ληφθεί μια απόφαση, έχει ληφθεί, τελείωσε, υπάρχει. Και πρέπει να ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία. Οπότε, το να προβλέψουμε επιπλέον ελαστικότητα, ευελιξία, είναι κάτι ασυνήθιστο. Μπορεί να είναι ενδιαφέρον, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει γίνει ποτέ νομίζω. Πάντως να τη συζητήσουμε. Να ελέγξουμε τη δυνατότητα αυτή. Μήπως μπορεί να υπάρχει τέτοια ευελιξία. Θα είναι βέβαια κάτι καινούριο στο ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά και στο διεθνές δίκαιο νομίζω. Να, λέει ο Πρόεδρος, μια νέα πρόκληση για τον εισηγητή. Τώρα, η κυρία Τούρνου και ο κύριος Τριανταφυλλίδης και μετά η κυρία Σαλτεμόσα. Έτσι, αυτή είναι η επόμενη τρεις. Ευχαριστώ για την τόσο ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας σήμερα που πραγματικά μας έδωσε νέες ιδέες. Δεν είναι μυστικό ότι πρόκειται για μια δύσκολη οδηγία και ότι έχουν ακουστεί πολλές επικρίσεις και από εδώ και από το Συμβούλιο και από τους καταναλωτές αλλά και από τις επιχειρήσεις. Το έχω μάθει αυτό. Και, και εμείς και εκείνοι μιλάμε για την μείωση της προστασίας του καταναλωτή. Αυτή είναι η ανησυχία μας. Όπως επίσης και η νομική αβεβαιότητα που καλύπτει αυτή την οδηγία. Εσείς μας δώσατε κάποιες νέες προοπτικές και σας ευχαριστώ ειλικρινά πολύ. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την βούληση που δείχνετε στην προσέγγιση της νομοθεσίας. Δεύτερον, επειδή είσαστε πιο ξεκάθαροι για το τι μπορεί να εναρμονιστεί και τι δεν μπορεί να αναρμονιστεί. Ήταν ε, ιδιαίτερα ακριβή αυτά που μας είπατε. Τώρα έχω κάποιες ερωτήσεις. Πρώτον, αν λέτε ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στην εναρμόνιση γιατί να μην διαγράψουμε το άρθρο 4. Επαναλαμβάνω, είναι ένα σαφές μήνυμα. Να έχουμε μια γενική προσέγγιση και μετά κατά βήμα να δούμε τι εναρμόζουμε. Άρθρο 4 λοιπόν. Αναφερθήκατε και εσείς σύντομα σε αυτό. Δεύτερον, τι ιδέα έχετε για να λυθούν τα νομικά ζητήματα που γύρονται όσον αφορά το εύρος εφαρμογής και τρίτον αναφερθήκατε, να κάτι καινούριο πάλι σήμερα, την, ε, τις εξαποστάσεως εμπορικές συναλλαγές και τις ε, απευθείας. Θα μπορούσατε να επεκταθείτε περισσότερο στις δυσκολίες. Αν έχουμε δύο διαφορετικά καθεστώτα, τι έχουμε να κερδίσουμε, αλλά κυρίως τι έχουμε να χάσουμε από μια τέτοια προσέγγιση. Υπάρχουν κάποια αρνητικά. Έπειτα, τι άλλες πρωτοβουλίες θα μπορούσαμε να περιλάβουμε, να συμπεριλάβουμε για την προστασία του καταναλωτή πέραν από αυτές που ήδη υπάρχουν. Που θα ήταν ίσως η ευθύνη του παραγωγού. Να, μια ιδέα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ την Επίτροπο για τις απαντήσεις που έχει δώσει, ιδιαίτερα στο θέμα της εναρμόνισης. Θα χαρόμουν πολύ αν μπορούσε να γίνει αυτό που είχε πει για την πλήρη εναρμόνιση στο ανώτατο επίπεδο. Αλλά έστω και αν αυτό δεν μπορεί να γίνει, θα συμφωνούσα πλήρως με την κυρία Γκέμπαρτ ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε οτιδήποτε που θα έχει ως αντίκτυπο την υποβάθμιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών δηλαδή η πλήρης εναρμόνιση εκεί όπου καταλήγει στην υποβάθμιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών μας είναι εντελώς απαράδεκτη. Ε, θέλω να αναφέρω κάτι για το θέμα των εγγύσεων στο κεφάλαιο 4. Εδώ υπάρχει μια αδυναμία στη μεταβίβαση των εγγύσεων. Οι εγγύησει συνοδεύουν το προϊόν και όχι τον αγοραστή. Ε, νομίζει η Επίτροπος ότι θα μπορούσε η Επιτροπή να εξετάσει αυτό το ζήτημα και να προσπαθήσει να το αλλάξει, γιατί μου φαίνεται λογικό οι εγγυήσει να είναι μεταβιβάσιμες ε, και να συνοδεύουν τον αγοραστή και όχι το προϊόν. Ευχαριστώ. Uh, thank you. Uh, Mrs. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ και την Επίτροπο βεβαίως. Νομίζω ότι ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον να την ακούσουμε σήμερα εδώ. Νομίζω επίσης ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι ήρθε εδώ για να συζητήσει μαζί μας όσον αφορά τις εξελίξεις ε, για τις οδηγίες αυτής. Όμως, πρέπει να παραδεχτούμε ότι ε, περνάω από τη μία αίσθηση στην άλλη, από το κρύο στο ζεστό. Δηλαδή, μία στιγμή μου φαίνεται ότι όλα πάνε πάρα πολύ καλά και τι ωραία είναι αυτά που ακούμε και μετά αμέσω μία ψυχρολουσία, όχι δεν είναι ακριβώ αυτό που θα θέλαμε. Και έχω την αίσθηση ότι τελικά θα χάσει, ε, την ίδια αίσθηση θα έχει ο καταναλωτή. δηλαδή θα χάσει και αυτός ε, την εμπιστοσύνη του. Τη μία φορά θα λέει «Α, πάρα πολύ ωραία είναι όλα αυτά» και την άλλη φορά θα αισθάνεται ασάφεια. Επομένω θα πρέπει να να θέσουμε κάποιες ε, προτεραιότητες. Ε, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σαφείς. Να δούμε δηλαδή ακριβώς πώς θα έχουν τα πράγματα για τους πολίτες και για τους καταναλωτές μετά από την οδηγία αυτή. Βεβαίως θεωρώ πάρα πολύ σημαντική την επιθυμία που έχετε, τη βούληση που έχετε ε, για συζήτηση. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αλλάξουν αρκετά πράγματα στην οδηγία και θα μπορούσαμε ενδεχομένως να δούμε ξεχωριστά οτιδήποτε ε, σχετίζεται με τις ε, διασυνοριακές ε, συναλλαγές. Ίσως θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε λοιπόν βήμα προς βήμα και να λύσουμε ένα-ένα τα προβλήματα. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Επίτροπε. Ήδη σαφώς είπα στην ε, εισαγωγική μου ομιλία ότι δεν πιστεύω ότι η υψηλότερη προστασία του καταναλωτή ε, μπορεί να αντιταχθεί ε, εις την εμπορική επιτυχία των επιχειρήσεων. Εγώ πιστεύω ότι η ε, καλύτερη αντιμετώπιση των ε, δικαιωμάτων των καταναλωτών θα δημιουργήσει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο καταναλωτικό κοινό και αυτό θα έχει καλά αποτελέσματα στην επιχειρηματικότητα. Όμως θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι πρέπει να προχωρήσουμε προς τα εμπρός ε, στην εσωτερική αγορά ενδυναμώνοντας την ασφάλεια και την ασφάλεια δικαίου ε, και την συνοχή ε, δικαίου όσον αφορά τις διασυνοριακές συναλλαγές. Και αυτό θα είναι καλό και για τον επιχειρηματικό κόσμο και για, τις, για τους καταναλωτές. Για τον επιχειρηματικό κόσμο ε, θα είναι καλό να μην έχουν 20, 30, 50 διαφορετικά συστήματα να εφαρμόσουν. Εάν έχουμε προστασία διασυνοριακών συναλλαγών, αυτό ταυτοχρόνως θα αποτελέσει κίνητρο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπουν σε αυτό το τομέα των διασυνοριακών πωλήσεων. Το άρθρο 4 φαίνεται ότι αποτελεί πρόβλημα για την σοσιαλιστική ομάδα. Αυτό είναι το, το κέντρο ενδιαφέροντος. Μπορώ να το καταλάβω βεβαίως. Όμως έχω πει επανειλημμένα ότι δεν θα επιμείνω σε πλήρη εναρμόνιση παντού. Έχω αναλύσει τα στοιχεία σε πέντε ομάδες και λέω ας πούμε ότι όσον αφορά τους ορισμούς π.χ. μπορεί να υπάρξει πλήρης εναρμόνισης και θα, ήταν, ε, θα είχε θετικό αποτέλεσμα ενώ πλήρης εναρμόνιση σε κάποιους άλλους τομείς ενδεχομένως ε, να μην ε, είναι απολύτως απαραίτητη ε, και αυτό, και απαντώ εδώ και στην κυρία Γκέμπχαρτ, ότι με τον τρόπο αυτό θα τροποποιείται το ε, άρθρο 4. Γιατί στην ουσία η πλήρης εναρμόνιση δεν αντιτίθεται εις ε, την προστασία των καταναλωτών στις περιπτώσεις που θα έχουμε πλήρη εναρμόνιση και στις άλλες περιπτώσεις σαφέστατα δεν προχωρούμε σε απολύτως πλήρη εναρμόνιση. Τώρα, το να ε, εφαρμόσουμε την οδηγία αυτή μονάχα σε μία κατηγορία συναλλαγών, ναι, ενδεχομένως. Δεν θα ήταν βεβαίως τόσο μακρόπνοη όσο ε, αυτή που έχουμε εδώ μπροστά μας, αλλά θα μπορούσε να αποτελέσει μία λύση. Ε, κοιτάξτε, εδώ κάνουμε μία ανοιχτή συζήτηση για τη βέλτιστη λύση. Αν αυτή είναι η βέλτιστη λύση, τότε θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να συμφωνήσει με την κατεύθυνση αυτή. Εγώ δεν θέλω να κλείσω καμία πόρτα και δεν θέλω να αποκλείσω κανένα ενδεχόμενο. Είναι γεγονός ότι έχω ξανασκεφτεί λίγο αυτά τα οποία είπα στην ε, ακρόαση επί τη βάση των όσων άκουσα και επομένως ε, θεωρώ ότι εάν κρατήσουμε μία άκαμπτη στάση δεν θα είναι εύκολο να εξαιρεθεί διέξοδος. Ο νομοθέτης δηλαδή δεν θα, ε, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να βρει ε, μία διέξοδο. Τώρα, μπορώ να εγγυηθώ ότι οι καταναλωτές δεν θα χάσουν δικαιώματα. Έχω την καλύτερη εγγύηση μπροστά μου. Γιατί δεν πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο θα συμφωνήσει με οτιδήποτε οδηγεί σε απώλεια των δικαιωμάτων των πολιτών. Ε, και αν το Κοινοβούλιο προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση, τότε θα έχει έρθει ο κόσμος ανάποδα. Και εγώ δεν θα καταλαβαίνω πλέον το ρόλο του Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι εσείς, σαν εκλεγμένοι εκπρόσωποι των πολιτών, παίζετε και θα συνεχίσετε να παίξετε τον ρόλο που σας αρμόζει και επομένως θα προστατέψετε τα δικαιώματα των πολιτών και των καταναλωτών. Σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Τριανταφυλλίδης για τις εγγυήσεις που πρέπει να, να ακολουθούν το προϊόν και όχι τον αγοραστή. Ναι, προφανώς συμβαίνει αυτό. Όμως, εάν το προϊόν αλλάζει χέρια από τον έναν αγοραστή στον άλλον, θα πρέπει να ακολουθεί και η εγγύηση. Είναι ένα πάρα πολύ μπερδεμένο περίπλοκο ζήτημα. Και εδώ σας κάνω μία έκκληση. Ας προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις που μπορεί να καταλάβει ο καταναλωτής. Πιστεύω ότι στο τέλος μπορεί να υπάρξει οδηγία προστασίας του καταναλωτή. Και τότε όλοι μας θα έχουμε παίξει καλά τον ρόλο μας όσον αφορά την σωστή επικοινωνία με τους ε, καταναλωτές. Θα έχουμε δηλαδή δώσει στους καταναλωτές να καταλάβουν κάποια πράγματα. Θα τους έχουμε εξηγήσει σωστά κάποια πράγματα. Όμως ε, θα πρέπει πάντα να έχουμε στο νου μας να μην βαραίνουμε πάρα πολύ τη βάρκα γιατί στο τέλος θα βυθιστεί. Χρειαζόμαστε τη βάρκα αυτή. Ας μην τη βαρύνουμε. Και όσο γίνεται, σας παρακαλώ, να διατηρήσουμε ε, ε, εύκολα κατανοητούς τους κανονισμούς. Τώρα, εάν περιοριστούμε μόνο στις διασυνοριακές συναλλαγές, βεβαίως θα είναι μία λύση μακράν της επιθυμητής, αλλά εάν το Κοινοβούλιο θεωρήσει ότι αυτή είναι η καλύτερη λύση, τότε θα προσπαθήσω κι εγώ να πείσω τους υπόλοιπους 26 επιτρόπους ότι αυτό είναι ο καλύτερος ε, δρο... η καλύτερη οδός διαφυγής. Πρόεδρος, θα δώσω το λόγο ε, στον εισηγητή στο τέλος. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο λοιπόν, γι' αυτό θα ήθελα οι ερωτήσεις των παρεμβενόντων να είναι σύντομες, έτσι ώστε να μπορέσει και η κυρία Επίτροπος να απαντήσει σε όλες. Τέσσερις ερωτήσεις λοιπόν, en bloc. Θα σας δώσουμε ένα ρολόι να το βλέπετε έτσι ώστε να μην μακρηγορήσετε. Ερωτήσεις ενό λεπτού αν είναι δυνατόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ ε, την, ε, ε, την εισηγήτρια. Θα χρησιμοποιήσω τη γλώσσα μου και δεν θα με ενοχλήσει αν δεν απαντήσετε εσείς ρωμανικά. <laughs> Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ε, μας εκφράζεται την άποψη της νέας Επιτροπής και χαιρόμαστε γιατί εδώ ε, βλέπουμε την εικόνα μιας ευέλικτης Επιτροπής και αυτό είναι σημαντικό. Χρειαζόμαστε βεβαίως ενιαίο πλαίσιο Χρειαζόμαστε όμως και ένα κανονιστικό πλαίσιο το οποίο θα είναι εύκολα κατανοητό από τους πολίτες και από την άλλη πλευρά βεβαίως δεν υπάρχει κανένας λόγος ένα ε, καταναλωτής ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο να χαίρει περισσότερων δικαιωμάτων από ότι ένα καταναλωτή ε, στη Βουλγαρία ή στην Ρουμανία. Επίσης θέλουμε να υπάρχει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που θα δίνει τα ίδια δικαιώματα στου καταναλωτέ των παλαιών και των νέων χωρών. Ε, πιστεύουμε ότι το, κοινο... Ε, ότι το Συμβούλιο και οι Κομισιόν πολλά μπορούν ε, να κάνουν και να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα τα οποία είναι πιο λεπτά για μας εδώ στο Κοινοβούλιο. Εάν προχωρήσουμε σε πλήρη εναρμόνιση ε, ε, θα, δοθεί η δυνατότητα ενδεχομένως σε κάποιες χώρες ε, να δημιουργήσουν επιπλέον νομοθετικά πλαίσια, επιπλέον προστασία. Τέλος, να σχολιάσω αυτά που είπατε σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εκστρατεία. Να σας πω ότι εμείς στην πολιτική μου ομάδα αποφασίσαμε ότι θα ξεκινήσουμε μια εκστρατεία πληροφόρησης όσον αφορά την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στις χώρες μας ε, και ε, βεβαίως θα κάνουμε και μια εκστρατεία για την ενιαία αγορά. Ε, θα μιλήσω στη γλώσσα μου εάν συμφωνείτε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο και σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ βασικά. Συγχρόνως όμως θέλω να υπογραμμίσω ότι δεν ξέρω κατά πόσο εδώ ψάχνουμε να βρούμε στόχους οι οποίοι να μην συμβιβάζονται. Τι θέλουμε. Θέλουμε πρώτα απ' όλα να προστατεύσουμε τους καταναλωτές. Και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος? Η οδηγία. Γι' αυτό και λέγεται οδηγία για την προστασία των καταναλωτών. Δεύτερο στόχος είναι πώς θα ενισχύσουμε το διασυνοριακό εμπόριο. Πιστεύω ότι η οδηγία για την προστασία των καταναλωτών προσπαθεί να πετύχει και τους δύο στόχους συγχρόνως. Πιστεύοντας ότι για να έχουμε αποτελέσματα προς τη μία κατεύθυνση πρέπει να έχουμε αποτελέσματα και προς την άλλη κατεύθυνση. Αυτό όμως είναι το πρόβλημα που μας δυσκολεύει και μας δημιουργεί τόσες δυσκολίες. Τι γίνεται με τον ΦΠΑ, τι γίνεται με την πληρωμή σε ρευστό όταν παραδίδεται το εμπόρευμα. Τι γίνεται με την εγγύηση όταν πρόκειται για πιστοτικές κάρτες κάποιος ο οποίος δίνει το όνομά του και τον αριθμό της πιστητικής του κάρτας. Πώς μπορούμε να έχουμε την εγγύηση ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί, δεν θα υπάρξει κατάχρηση. Αυτά είναι προβλήματα τα οποία ξέρω ότι δεν μπορείτε μόνοι σας να τα λύσετε. Χρειάζεται συνεργασία και με άλλου επιτρόπους. Πάντως, κύριε Επίτροπε, εσείς δείξατε, επιδείξατε πνεύμα συμβιβαστικό και μας προτείνατε να χωρίσουμε τις δύο πραγματικότητες, τις δύο καταστάσεις. Από τη μία το εμπόριο το οποίο ίσω σύστομα face to face, το άμεσο, η άμεση εμπορική συναλλαγή και από την άλλη μεριά χωριστά να έχουμε τις συναλλαγές εξ αποστάσεως. Και ότι έτσι μπορεί να υπάρχει διαφορετική συμπεριφορά. Αλλά τότε δεν κινδυνεύουμε να καταλήξουμε σε δύο νομοθεσίες οι οποίες μπορεί να είναι και αντιφατικές μερικές φορές μεταξύ τους. Ευχαριστώ. Uh, thank you very much, um, Ευχαριστώ. Κύριε Στάλλαρ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ την Επίτροπο. Πολλά ακούστηκαν, δεν θα τα επαναλάβω. Αλλά ήθελα να μιλήσω λίγο για τις εμπορικές συναλλαγές online. Και αν κάποιος αγοράσει ένα βιβλίο από το Amazon, ε, διαφέρει πάρα πολύ από το αν αγοράσει ένα μπάνιο. Θα πρέπει λοιπόν κάπως να βάλουμε κατηγορίες συναλλαγών και ποσά και την ίδια ώρα να κατηγοροποιήσουμε και τις επιχειρήσεις, μικρομεσαίες, μεγάλες πολυεθνικές. Θέλω λοιπόν να μπούμε λίγο σε κάποιες λεπτομέρειες και τύπους συναλλαγών. Το κόστος ε, διαφέρει πάρα πολύ. Όσον αφορά την πρόσβαση, μιλάμε για άμεσες συναλλαγές, face to face και μέσω διαδικτύου. Η πρόσβαση λοιπόν είναι πολύ σημαντική και η ασφάλεια, η προστασία. Λέτε ότι μόνο το 20% των καταναλωτών των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης νιώθουν ασφάλεια όταν συναλλάσσονται online. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να δούμε και όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την προστασία, με την ασφάλεια. Για όλες αυτές τις ε, συναλλαγές και πρέπει να προσέξουμε έτσι ώστε όπως αυξάνεται ο αριθμός αυτών των συναλλαγών μέσω διαδικτύου να μην ασφάνεται, να αυξάνεται συγγνώμη, και η ανασφάλεια. Πιστεύω λοιπόν ότι όλα αυτά θα πρέπει να τα σκεφτούμε προσεκτικά. Ευχαριστώ πολύ. Η Μπερναντέτ. Ευχαριστώ την Επίτροπο που είναι σήμερα μαζί μας. Σας είδαμε και στην προηγούμενη θητεία σας ότι πραγματικά σας αφορά το θέμα της προστασίας του καταναλωτή. Λέτε ότι ένας καταναλωτής που νιώθει ασφαλής, που έχει εμπιστοσύνη στην οικονομία, καταναλώνει καλύτερα και περισσότερο. Και αυτό είναι καλό και για την εσωτερική αγορά, αλλά και για την οικονομία της Ευρώπης. Η αναρμόνιση λοιπόν θα πρέπει να είναι μια αναρμόνιση στόχευμένη έτσι ώστε αυτοί που έχουν χαμηλή προστασία του καταναλωτή να ανυψώσουν το επίπεδο, αυτοί όμως που έχουν υψηλή προστασία να μπορέσουν να την διατηρήσουν. Μιλήσατε για την ενημέρωση και για την προσυμβατική ενημέρωση και πληροφορία που δίνουμε στον καταναλωτή. Έχετε δίκιο. Θα πρέπει να έχουμε μία πλήρη ενημέρωση και πληροφόρηση των καταναλωτών πριν συνάψουν μια συμφωνία και να υπάρξει νομική ασφάλεια. Πρέπει επίσης να ξαναδούμε τις προθεσμίες για να αποφασίσει κανείς ε, την εμπορική συναλλαγή. Επίσης να υπάρχει και μία χρονική περίοδος μετά την απόφαση αυτή έτσι ώστε να μπορέσει να αλλάξει γνώμη ενδεχομένως ο καταναλωτής, έτσι ώστε να μειώσουμε τους κινδύνους και να προστατεύσουμε περισσότερο τους καταναλωτές. Σας κάνω επίσης και μια άμεση ερώτηση. Όσον αφορά τις απάτες αυτές τις συναλλαγές online, ποια είναι η άποψή σας και πώς μπορούμε να κάνουμε συλλογικές προσφυγές όπως προβλέπει ο Ευρωπαϊκός νόμος και όχι όπως προβλέπει ε, ο Αμερικανικός. Η Επίτροπος. η πλήρης εναρμόνιση πιστεύω ότι δεν θα περάσει. Πραγματικά βλέπω τις πλειοψηφίες και εδώ στο Κοινοβούλιο αλλά και στο Συμβούλιο. Η πλήρης εναρμόνιση δεν θα προχωρήσει. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε λύση. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς σας λέω ότι είμαι διατηθμένη να ακολουθήσω το Κοινοβούλιο και, την, ε, και το Συμβούλιο σε άλλες κατευθύνσεις. Η ενημέρωση είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά όταν ολοκληρωθεί θα πρέπει να βρούμε λύσεις και να τις επιλέξουμε και να τις εφαρμόσουμε. Οι στόχοι είναι τελείως διαφορετικοί εδώ, η μεν και η δε. Εγώ δεν είμαι σίγουρη. Κοιτάξτε παραδείγματο χάρη, η περιαγωγή. Μας είπαν οι επιχειρήσεις ότι θα φαλυρίσουν εάν πιέσουμε όσον αφορά ε, το θέμα της περιαγωγής. Τελικά, τι είδαμε τον πρώτο χρόνο, οι καταναλωτές χρησιμοποίησαν τα κινητά τους 30% παραπάνω από ότι το προηγούμενο χρόνο. Άρα τι έγινε. Η κατανάλωση αυξήθηκε δραστικά. Και αυτό πραγματικά με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στον κόσμο του διαδικτύου, αν υπάρχει περισσότερη ασφάλεια, περισσότερη νομική ασφάλεια και για τις επιχειρήσεις και για τον καταναλωτή, το εμπόριο, ο όγκος των συναλλαγών, η κατανάλωση θα αυξηθεί. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να το δοκιμάσουμε. Το πολύ χαμηλό ποσοστό που βλέπουμε σήμερα στην Ευρώπη είναι μια χαμένη ευκαιρία και για τους καταναλωτές και για τις εταιρείες. Βεβαίως θα χρειαστούμε τη βοήθεια και άλλων επιτρόπων. Και φυσικά και οι 26 άλλοι επίτροποι θα πρέπει να αποφανθούν. Άλλοι πολύ, άλλοι λίγο. Αλλά σαφώς και πρόκειται για μια συλλογική απόφαση της Επιτροπής. Και ο κίνδυνος όσον αφορά τη διαφοροποίηση μεταξύ των εμπορικών συναλλαγών που θα διέπουν τις face-to-face -face to face συναλλαγες τις άμεσες συναλλαγές και τις συναλλαγές τις ηλεκτρονικές, είναι επικίνδυνες. Βεβαίως και θέλουμε εναρμόνιση περισσότερη, αλλά προχωράμε σιγά-σιγά προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι όριμο το θέμα για πλήρη αναμόνιση σήμερα, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε και τις επιλογές μας. Και θα ήθελα να πω στην κυρία Στάιλερ ότι βεβαίως υπάρχουν διαφορετικές συναλλαγές. Ακόμα και στις άμεσες συναλλαγές, στις face-to-face, -face, υπάρχουν κατηγορίες συναλλαγών. Εάν παραδείγματος χάρη Διότι όπως ξέρουμε σήμερα είναι εύκολο να αγοράσει κανείς ένα τραγούδι στο διαδίκτυο. Ξέρετε όμως ότι αν ένας νέος προσπαθήσει να αγοράσει νόμιμα ένα τραγούδι δύο-τρεις φορές και αποτύχει, θα το κάνει παράνομα. Θα πρέπει λοιπόν να παρακολουθήσουμε αυτές τις εξελίξεις και να βρούμε ασφαλείς τρόπους έτσι ώστε να δημιουργήσουμε στο διαδίκτυο ασφαλείς, νόμιμες και εύκολες διαδικασίες. Όπως είπε και η κυρία Βέρνιο, πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να αναλαμβάνουν τον κίνδυνο μιας απάτης οι καταναλωτές και ότι θα πρέπει να θεσπίσουμε σαφείς διαδικασίες προσφυγής, ακόμα και αν αυτές είναι συλλογικές, ομαδικές προσφυγές. Τέλος τώρα δεν μιλάω σαν επίτροπος, μιλάω σαν Vivian Redding. Και αυτές οι ομαδικές προσφυγές τελικά θα μας οδηγήσουν σε ένα αμερικάνικο σύστημα και αυτό βέβαια είναι καταστροφική συνέπεια. Ξέρω ότι δεν είστε υπέρ. Γι' αυτό και εγώ είμαι πολύ επιφυλακτική εξάλλου. Η συζήτηση, εν πάση περιπτώσει, συνεχίζεται στην Επιτροπή για το θέμα αυτό. Υπάρχουν επίτροποι που είναι αρμόδιοι για το θέμα και πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει ακόμα απόφαση. Γι' αυτό και είμαι τόσο προσεκτική ε, και εκφράζω μόνο την προσωπική μου ε, γνώμη. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Ράπτη, η κυρία Ρούλε και ο κύριος Άριας. Έχετε το λόγο. Έχετε ένα λεπτό. Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, καλώς ήρθατε. Μου αρέσει ο τρόπος που εργάζεστε σας θυμάμαι από την Ελλάδα όταν ήσασταν ξανά επίτροπος με σοσιαλιστική κυβέρνηση στην Ελλάδα και Υπουργό Παιδείας στον κύριο Ευθυμίου που έχει υπάρξει και Ευρωβουλευτής. Ε, θέλω να σας πω μια σκέψη μου. Η σκέψη μου είναι η εξής. Χτες ήταν η Παγκόσμια ημέρα των καταναλωτών. Η οδηγία αναφέρεται στους καταναλωτές. Ωστόσο στην ομιλία σας χθες στη Μαδρίτη όπως είδα, αναφερθήκατε πρώτα στις επιχειρήσεις. Όλη η συζήτηση που γίνεται εδώ, όλη αυτή την ώρα, πάντα ξεκινάει για το καλό των καταναλωτών, αλλά καταλήγουμε στις επιχειρήσεις. Και πραγματικά ξέροντας και πάλι ε, υπογραμμίζω τον τρόπο που εργάζεστε και το πόσο μεθοδικοί είστε, ε, θα ήθελα να με πείσετε για το ότι η προτεραιότητά σας είναι οι καταναλωτές. Είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. και εγώ θα προσπαθήσω να είμαι πολύ πολύ σύντομη. Σας ευχαριστώ πολύ για τις προτάσεις σας και για τις πολύ ρεαλιστικές σας, αν θέλετε, θέσεις και προσεγγίσεις. Σας ευχαριστώ πολύ όσον αφορά τους ορισμούς. Συμφωνώ και εγώ μαζί σας ότι θα πρέπει πραγματικά οι ορισμοί να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Έχω και μία ερώτηση. Κατάλαβα καλά ότι θα υποστηρίξετε την αλλαγή του άρθρου 4. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το ξέρουμε. Και μιλήσατε για μια σταδιακή προσέγγιση. Έχει νόημα αυτή. Όσον αφορά τις εμπορικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου, το θέμα των πληρωμών και το θέμα της προστασίας των δεδομένων είναι ίσως το πιο σημαντικό, γιατί μόνο τότε θα αυξηθεί ο αριθμός των συναλλαγών στο διαδίκτυο. Ο κύριος Άριας είναι ο τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρία Ρέντινγκ, σας ευχαριστούμε πολύ για τα σχόλιά σας και για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Συμφωνώ απολύτως με τις θέσεις σας όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο. Βεβαίως αυτό αφορά άμεσα τα δικαιώματα των καταναλωτών και ίσως θα μπορούσαμε εδώ να πούμε με σαφή τρόπο ότι πραγματικά πιστεύουμε, έχουμε εμπιστοσύνη στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά και να εξηγήσουμε και στους καταναλωτές αλλά και στους εκλογείς μας τελικά ότι θα τους προστατεύσουμε, θα ασχοληθούμε πραγματικά με τα δικαιώματά τους. Σε μία από τις απαντήσεις που δώσατε μιλήσατε για την υπερβολή όσον αφορά τα δικαιώματα. Την υπερβολική δόση, αν θέλετε, των δικαιωμάτων που πολλές φορές προκαλούν σύγχυση στους καταναλωτές. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να γίνουν γνωστά τα δικαιώματα των καταναλωτών, καταρχήν βάσει της νομοθεσίας της εθνικής. Παραδείγματος χάρη, εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι οι Ισπανοί καταναλωτές γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και σαφώς και δεν είμαι υπέρ της πλήρους εναρμόνισης, γιατί κάποιοι καταναλωτές θα πληγούν, θα υποβαθμιστεί η προστασία τους το επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων τους. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξής. Πώς μπορούμε να εναρμονίσουμε προς τα πάνω για 27 χώρες βάσει της οδηγίας την οποία επεξεργαζόμαστε. Πρέπει να δείξουμε δημιουργικότητα και ακρίβεια σε κάποια πολύ συγκεκριμένα σημεία γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια κάποια εναρμόνιση. Ευχαριστώ πολύ η Επίτροπος και κατόπιν ο Ανδρέας Φαμπ, ο οποίος θα μας παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο θέλει να προχωρήσει από εδώ και πέρα. Έχετε το λόγο. Κυρία Ράπτη, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να είμαστε υπέρ των καταναλωτών, άρα κατά των επιχειρήσεων ή υπέρ των επιχειρήσεων, άρα κατά των καταναλωτών. Πραγματικά πιστεύω ότι η πολιτική μας πρέπει να βασίζεται σε σαφείς κανόνες για όλους. Και αν καταλάβατε αυτά που πρεσβεύω και επειδή πρόκειται για μια οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν υπάρχει απόλυτη, αν θέλετε, υπεροχή των δικαιωμάτων του καταναλωτή. Θα πρέπει να βρούμε την βέλτιστη, αν θέλετε, προστασία. Την βέλτιστη, όχι τη μέγιστη, την βέλτιστη. Κάτι που επιτρέπει την νομική ασφάλεια για τις εταιρείε, για τις επιχειρήσεις. Γι' αυτό και όταν μιλάω για επιχειρήσεις θέλω να κατανοήσετε ότι μιλάω κυρίως για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μεγάλες πολυεθνικές δεν έχουν πρόβλημα. Οι μικρομεσαίες όμως επιχειρήσεις, κυρίως αυτές που εργάζονται παραδείγματος χάρη σε, συνοριακές, ε, σε συνοριακές περιοχές όπως το Λουξεμβούργο που γνωρίζω καλά. Εκεί θα πρέπει πραγματικά να αποφύγουμε στρέβλωση ανταγωνισμού. Και είναι οικονομικό το θέμα από εκεί και πέρα βεβαίως. Πρέπει, οφείλουμε να δημιουργήσουμε ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι οι δραστηριότητες όσον αφορά την κατανάλωση που προστατεύουν τα δικαιώματα μπορούν να ενισχύσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αν αυτά γίνουν με λογική και με ισορροπημένο τρόπο. Δεν είναι θέμα λοιπόν προτεραιότητας. Εδώ μιλάμε για τα δικαιώματα των καταναλωτών, αλλά δεν πρέπει τα δικαιώματα των καταναλωτών να είναι εις βάρος της ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γιατί θα κλείσουν, θα χάσουμε ανάπτυξη, θα χάσουμε θέσεις απασχόλησης και αυτό είναι το ζητούμενο. Κυρία Ρίλα, είναι σαφές αυτό που είπα. Το άρθρο 4 αν τελικά το εξαλείψουμε, αν δηλαδή τελικά το Κοινοβούλιο δεν θέλει πλήρη εναρμόνιση, να το σβήσουμε το άρθρο 4. Και πρέπει να δούμε εδώ τι θα μπει μέσα στους διάφορους ορισμούς. Το άρθρο 4, δεν θέλω να μιλήσω ιδεολογικά αν θέλετε. Πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο 4, διότι αφού δεν δεχόμαστε την πλήρη εναρμόνιση πρέπει να τροποποιήσουμε το άρθρο 4. Η πλήρη εναρμόνιση αν εξαλειφθεί τελείω, θα εξαλειφθεί και το άρθρο 4. Αλλά αυτό θα γίνει στο τέλο τη διαδικασία. Α ξεκινήσουμε με την επίλυση των επιμέρου προβλημάτων και σιγά σιγά θα φτάσουμε και στην ιδεολογία, στι βασικέ και θεμελιώδει αρχέ του κειμένου συμφωνώ απόλυτα όταν λέτε ότι πρέπει να βρούμε λύσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Εγώ είμαι άκαμπτη επ' αυτού. Και βεβαίως οι καταναλωτές δεν πρόκειται να νιώθουν καμία εμπιστοσύνη όταν συναλλάσσονται στο διαδίκτυο εάν η ασφάλεια των πληρωμών δεν είναι εγγυημένη. Αυτό είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Η κυρία Κρούς πραγματικά θα πρέπει να εργαστεί σκληρά για τον τομέα αυτό. Η εμπιστοσύνη είναι θεμελιώδης αρχή. Αν ο καταναλωτής νιώθει ασφαλής, ότι η πληρωμή θα γίνει με ασφαλή τρόπο, ότι θα λάβει το προϊόν που παράγγειλε και πλήρωσε εγκαίρος και σε καλή κατάσταση, θα αγοράζει περισσότερο στο διαδίκτυο. Εάν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πολλούν μέσω του διαδικτύου είναι σίγουροι ότι οι πληρωμές θα φτάσουν, θα αυξηθούν οι πληρωμές αυτές. Σήμερα το 60% των μη εξοφλημένων συναλλαγών στο διαδίκτυο δεν πληρώνονται. Δεν υπάρχει τρόπος προσφυγής και πληρωμής έστω καθυστερημένης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό δημιουργεί μια μεγάλη ανασφάλεια και θα πρέπει να συνεργαστούμε και με άλλους επιτρόπους έτσι ώστε να επιληφθούμε σφαιρικά του ζητήματος. Κύριε Αρίας, θα ήθελα με μαγικό τρόπο να σας πω ναι, αυξάνουμε την προστασία εν μία νυχτή. Αυτό θα ήταν τέλειο. Αλλά επειδή είμαι πολιτικός, σας λέω ότι αυτό δεν γίνεται. Και είμαι σίγουρη ότι θα φτάσουμε με τη βοήθεια του Κοινοβουλίου στο βέλτιστο σημείο. Το ελπίζω τουλάχιστον. Uh, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Επίτρεπε, καθότι υποβάλλατε νέες ιδέες, πολλές νέες ιδέες και δυνατότητες για λύσεις. Ο Ανδρέας Φαμπ πολύ σύντομα να μας παρουσιάσει τι θα κάνει από εδώ και πέρα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε. Έχω έξι σημεία και πολύ σύντομα θα σας τα παρουσιάσω. Πρώτον, ο συνάδελφος Οσφορ έφυγε δυστυχώς. Αναφέρθηκε στο θέμα της αξιολόγησης του αντικτύπου. Διαβάζω το κείμενό σας στα αγγλικά που λέει ότι πρέπει να αξιολογηθεί αυτό και αυτό και αυτό. Το θέμα λοιπόν είναι και το συζήτησαν σήμερα οι συντονιστές, τι έγγραφα, briefing papers θα πρέπει να προετοιμάσουμε για το θέμα αυτό. Δεύτερον, τα δικαιώματα των καταναλωτών και οι οργανώσεις προστασίας των καταναλωτών φοβούνται ότι οι λεγόμενοι μαύροι κατάλογοι, απαγορευτικοί κατάλογοι, blacklist, δυστυχώς παίρνουν λανθασμένη κατεύθυνση. Εσείς λοιπόν κύριε Επίτροπε θα πρέπει να μπορείτε να επιληφθείτε του θέματος και να πείτε ότι εδώ κάτι πρέπει να γίνει. Χρειαζόμαστε περισσότερη ευελιξία, περισσότερη πειθαρχία και γνώση της αγοράς. Τρίτο σημείο, η πλήρης εναρμόνιση. Εγώ θα ήθελα να ακούσουμε την συνάδελφο Τούρνερ, η οποία μίλησε για μία μηχανική αναπροσαρμογή και μία πλήρη εναρμόνιση η οποία ουσιαστικά αντιμετωπίζει σαν ένα άκαπτον σύνολο το θέμα. Θα πρέπει πραγματικά σταδιακά να προχωρήσουμε και σε αυτό νομίζω συμφωνείτε. Μιλήσατε επίσης για την ενημερωτική εκστρατεία. Είμαι πεπισμένος ότι όσο πιο διαφανή είναι τα δικαιώματα, τόσο πιο σοβαρά μπορεί ο καταναλωτής να τα πάρει υπόψη του και τόσο πιο εύκολα θα υλοποιηθούν και θα εφαρμοστούν στην πράξη. Η κυρία Βερνιό έχει δίκιο και αυτό είναι το πέμπτο μου σημείο ότι πολλές φορές δεν είναι εύκολο να γίνει να βρεθεί η διαχωριστική γραμμή μεταξύ αυτών των εξαποστάσεων συναλλαγών και των άλλων. Εγώ θα συνεχίσω να επεξεργάζομαι όλα αυτά τα σημεία και ελπίζω ότι μέχρι τις καλοκαιρινές διακοπές θα μπορώ να υποβάλω το σύνολο του κειμένου. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την κυρία Ρέντινγκ εκ μέρους της Επιτροπής μας που ήρθε και τόσο δυναμικά απάντησε στις ερωτήσεις μας και έκανε και κάποιες προτάσεις. Πιστεύω ότι προχωρήσαμε περισσότερο σήμερα το απόγευμα από ό,τι έχουμε προχωρήσει σε όλη τη συζήτηση από τότε που ξεκίνησε. Τώρα λοιπόν το μπαλάκι είναι στο δικό μας το γήπεδο. Θα τα ξαναπούμε πάντως όταν θα έχουμε και εμείς να προτείνουμε κάποιες λύσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε άλλο ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη. Γι' αυτό σας παρακαλώ όσοι καταλείπετε την αίθουσα ησύχω. Κύριε Ρέπο, μήπως να περιμένουμε τέσσερα λεπτάκια μέχρι να βγουν από την αίθουσα όσοι αποχωρούν.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 Παρακαλώ όσοι βγαίνετε από την αίθουσα να συνεχίσετε τα πηγαδάκια εκτός αιθούσης γιατί θέλω να προχωρήσουμε και να περάσουμε σε μια σημαντική γνωμοδότηση του συγγετή μας του κύριου Ρέπο για την κοινοτική πολιτική και την καινοτομία σε ένα μεταβελόμενο κόσμο. Έχουμε δέκα τροπολογίες, αυτή τη φορά είναι η δεύτερη που θα συζητήσουμε. Οπότε παρακαλώ τον εισηγητή να πάρει το λόγο, να μας πει ό,τι έχει να μας πει και να αντιδράσει στις τροπολογίες που έχουν ε, κατατεθεί μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πολύ, κυρίες και κύριοι. Ήταν πραγματικά καινοτόμο να ακούσουμε μια τόσο καινοτόμο επίτροπο, όπως παρουσιάστηκε εδώ σήμερα η κυρία Ρέντιν. Αλλά θέλω να πω πρώτα απ' όλα κάτι για τη στρατηγική του 2020. Ίσως να παρατηρήσατε ότι οι προτεραιότητες στη στρατηγική αυτή είναι μεταξύ άλλων ανάπτυξη στην ψηφιακή ατζέντα, στην εκπαίδευση. Ένας από τους στόχους της στρατηγικής είναι μια καινοτόμος ένωση. Έρευνα λοιπόν, καινοτομία, άρα τέτοιες πολιτικές πρέπει να έχουμε ως στόχο για το μέλλον. Πρέπει πρώτα απ' όλα να αποφασίσουμε για κοινούς στόχους και τι προκλήσεις καταρχήν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. Συντονισμένο όμως πρέπει να προχωρήσουμε και σε συνεργασία μεταξύ μας, γιατί έτσι θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Θέλουμε λοιπόν έναν ευρωπαϊκό χώρο καινοτομία. Αυτός είναι ο δρόμος, αυτό είναι το κλειδί. Η έρευνα και οι αγορές θα πρέπει να βρίσκονται πιο κοντά μεταξύ τους. Έτσι ώστε να δημιουργούνται τα προϊόντα τα οποία μας χρειάζονται, τα οποία, για τα οποία υπάρχει ζήτηση. Η καινοτομία έχει πολύ σημαντική θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το πρόβλημα με την καινοτομία είναι ότι δεν ξέρουμε πώς να υποφεληθούμε από τη γνώση, από τις πληροφορίες που έχουμε. Μια ιδέα καινοτομία είναι καλή στην αρχή της αλυσίδας. Μετά τι την κάνεις. Έχουμε λοιπόν πολλά ακόμα να κάνουμε. Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την καινοτομία πρέπει να έχουν πόρους για να προχωρήσουν. Πράγμα που μας φέρνει στην καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Πρέπει επίσης να αναπτύξουμε την ευρωπαϊκή πατέντα, η οποία θα προσφέρει στις επιχειρήσεις πολλά ευρώ. Όπως επίσης και θα βοηθήσει να εξοικονομήσουμε χρήματα Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια εναρμόνιση σε αυτό το τομέα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο δημόσιος τομέας είναι σημαντικός γιατί η κρατική χρηματοδότηση μπορεί να στηρίξει την καινοτομία. Όλοι έχουμε να μάθουμε από την εσωτερική αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών και τις πρακτικές που ακολουθούν εκεί. Για να διατηρηθεί η ευρωπαϊκή καινοτομία πρέπει τα οικονομικά μέσα να είναι πιο απλά και η διαχείρισή τους να είναι πιο απλή. Έρχομαι τώρα σε κάποια ακόμα σημεία, τα οποία αναφέρονται στο κείμενό μου. Δέκα τροπολογίες υποβλήθηκαν, για τις οποίες θέλω να ευχαριστήσω και την κυρία Βανόβα και τον κύριο Κρότσμαντ για τις τροπολογίες τους δεν μπορώ να πω ότι διαφωνώ ιδιαίτερα με τις τροπολογίες αυτές. Μπορώ να τις δεχτώ όλες. Εγώ ίδιος έχω υποβάλει δύο τροπολογίες μετά από τη συζήτηση που κάναμε την τελευταία φορά. Και για αυτές τις τροπολογίες τι έχω σκεφτεί. Έχω σκεφτεί ότι στο μέλλον η καινοτομία πρέπει να επικεντρώνεται στις ανάγκες του καταναλωτή και των κοινωνιών. Άρα λοιπόν η έρευνα και η καινοτομία πρέπει να ακολουθήσει την ζήτηση για καινοτομία. Ο χρήστης, ο καταναλωτής έχει δικαιώματα και πλεονεκτήματα τα οποία πρέπει να τηρήσουμε, να προστατεύσουμε. Στην άλλη μου τροπολογία μιλάω για την χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας. Ο κύριος Σβάρ στο δικό του το σημείο λέει ότι μόνο η Φιλανδία και η Σουηδία, μόνο δύο ευρωπαϊκές χώρες έχουν πάνω από 3% του ΑΕΠ για την καινοτομία. Και πάνω από 10 χώρες ε, δίνουν κάτω από 1% του ΑΕΠ στην έρευνα και την καινοτομία. Η χρηματοδότηση λοιπόν είναι πολύ σημαντική, ιδίω τώρα που είμαστε σε περίοδο κρίσης, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να προωθήσουμε την απασχόληση. Ο στόχος του 3% που τέθηκε στη Βαρκελόνη αποτελεί μέρος της στρατηγικής για το 2020. Αποτελεί δηλαδή έναν δίκτυ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριε Σιγητά, για τόσα πολύτιμα μας παρουσιάσετε. Εδώ έχουμε αναπληρωτέ νομίζω, όχι σκιώδεις. Δεν ξέρω για να δω ποιο θέλει το λόγο. Ο κύριος Σφαμπ ε, για την κυρία Ιβάνοβα, ο κύριος Κρότσμαν εδώ, ο κύριος Βίλον δεν είναι εδώ. Η κυρία Ρούλε θα μιλήσει... Κύριε Κρότσμαν, είσαστε σκιώδης. Πρώτα οι και μετά οι αναπληρωτές σκιώδεις. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι όντως σύντομος. Συμφωνώ με τις περισσότερες τροπολογίες και εγώ και πιστεύω πράγματι ότι στο θέμα της καινοτομίας πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με την εσωτερική αγορά. Το θέμα της ευρωπαϊκής πατέντας για μένα είναι στοιχείο κλειδί, γιατί μπορούμε να εξοικονομήσουμε πάρα πολλά χρήματα έχοντας ενιαίες διαδικασίες όσον αφορά την πατέντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν ένα ευρωπαϊκό σύστημα πατέντας χρειάζεται και ένα ευρωπαϊκό δικαστήριο για ό,τι διαφωνίες προκύπτουν σε θέματα πατέντας. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι οι τεχνολογίες ε, κλειδί πρέπει να προωθούνται μέσω δικών μας μηνυμάτων εκτός άλλων. Εμείς συμφωνούμε, αλλά όταν πρόκειται για την καινοτομία πρέπει να σκεφτόμαστε και θέματα όπως είναι η νανοτεχνολογία. Αλλά χωρίς να ξεχνάμε τους κινδύνους που μπορεί να ελοχεύει μια τέτοια τεχνολογία. Στα θέματα της έρευνας δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι χρειάζονται προδιαγραφές για τους ίδιους τους ερευνητές, για να μην τίθενται οι ίδιοι σε κίνδυνο. Πρέπει να αποφεληθούμε από ό,τι μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία. Μιλούσαμε για την αιωλική ενέργεια και λέγαμε ότι στο μέλλον αν τα μπορούν να χρησιμοποιήσουν νανοτεχνολογία μπορεί να είναι ε, αυτοκίνητα τα οποία θα καταναλώνουν αλλιώς ενέργεια. Θα χρησιμοποιούμε λέτε την νανοτεχνολογία για να φτιάξουμε ενέργεια. Όλα αυτά για να προωθήσουμε τις ενέργειες εκείνες οι οποίες αναδημιουργούνται, δεν χάνονται. Η κυρία Ρούλα. Ευχαριστώ. Δεν κατέθεσα εγώ τροπολογίες. Πριν μιλήσαμε για την τυποποίηση. Το θέμα της τυποποίησης πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό για την καινοτομία και δυστυχώς ξέχασα να υποβάλω τροπολογία. Ίσως θα μπορούσαμε κάπου να προσθέσουμε μισή πρόταση. Το λέω, το παραδέχομαι, το ξέχασα. Αλλά αυτή η ιδέα θα μπορούσε να προσθέσει πολλά. Κατά τα άλλα, η έκθεση είναι πάρα πολύ καλή. Πρόεδρος, αν συμφωνούν και οι συνάδελφοι, με μια προφορική τροπολογία μπορούμε να το πετύχουμε. Αύριο θα ψηφίσουμε, οπότε φροντίστε ακόμα σήμερα να το τακτοποιήσετε. Σφαμπ. Ευχαριστώ. Το επόμενο θέμα, το οποίο θέλω να θίξω εκ μέρους της κυρίας Ιβάνοβα Ιωπελίπη, είναι το εξή. Καταρχήν, η κυρία Ιβάνοβα, σας ευχαριστεί πολύ για την έκθεση που τη θεωρεί πολύ καλή. Δεύτερον, είπατε μόλις ότι συζητάμε την έρευνα και την καινοτομία και τι ξοδεύουν για αυτή οι διάφορες χώρες το κείμενο για το 2020 λέμε ότι θέλουμε το 3% αλλά δεν θα αρκεστούμε σε ένα έγγραφο. Λέμε ότι και σε εθνικό επίπεδο και στις 27 χώρες, όχι μόνο στη Σουηδία και στη Φιλανδία, παντού πρέπει να επιτευχθεί αυτό το 3%. Σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παλιότερα υπήρχαν χώρες όπως η Φιλανδία και η Σουηδία που ε, είχαν μεγαλύτερο ποσοστό και άλλε χώρε λέγανε δεν πειράζει, θα πετύχουμε το μέσο όρο αφού η Σουηδία και η Φιλανδία κάνουν καλύτερα πράγματα, εμεί μπορούμε να κάνουμε λιγότερα. Ε, όχι, δεν είναι έτσι. Υπάρχουν κάποιε τροπολογίε από την κυρία Ιβάνοβα. Στο άρθρο αριθμό 1... Εσείς μιλάτε για την σωστή, την εύρυθμη λειτουργία της ιστορικής αγοράς. Η κυρία Ιβάνοβα λέει ότι πρέπει να αναφέρονται εδώ οι μικρές και μεσέ επιχειρήσεις και ότι αυτές προωθούν την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Έπειτα, τροπολογία 9 για το ρόλο που παίζει η αγορά ε, χρησιμοποιώντας την ε, καινοτομία. Οι καταναλωτές λοιπόν πρέπει να έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν την καινοτομία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Απαλέτο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνο για την πολιτική καινοτομία. Θέλετε να σχολιάσετε παρακαλώ για την έκθεση του κυρίου Ρέπο ή ό,τι άλλο έχετε να μας πείτε πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Ρέπο για να κλείσουμε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομος. Όλα αυτά τα θέματα που αναφέρονται στην έκθεση ε, βρίσκουν σύμφωνη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χαιρόμαστε που έχουμε τη στήριξή σας αυτή, γιατί έτσι μπορούμε κι εμείς να προχωρήσουμε σε φιλόδοξες προτάσεις όσον αφορά την στρατηγική του 2020. Ευχαριστούμε. Κύριε Ρέπο, έχετε κάτι να πείτε. Αύριο στις 10 θα ψηφίσουμε την έκθεσή σας. Η κυρία Ρούλη είπε ότι έχει ένα σημείο, να δούμε πώς θα το συμπεριλάβουμε. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι όντως μπορούμε να φροντίσουμε για την προσθήκη αυτή της κυρίας Ρούλε. Μπορώ να το δεχτώ, ναι. Πρόεδρος, ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ένα πράγμα έχω να σας ζητήσω. Στην τελευταία σας τροπολογία, αριθμός 10, Μιλάτε για τη χρηματοδότηση της έρευνας και για τη διάθεση του 3% του ΕΠ. Νόμιζα ότι ήταν το σύνολο. Δεν ήταν μόνο η κυβερνητική δαπάνη, ήταν η συνολική δαπάνη. Είναι έτσι ή όχι. Γιατί λέτε ότι τα κράτη-μέλη να αυξήσουν τη χρηματοδότηση και τα λοιπά για να φτάσουν στο 3%. Μα μόνο για τα κράτη-μέλη μιλάμε ή και για ιδιωτικέ επενδύσει ενδεχομένω. Δεν ξέρω αν έχετε την απάντηση τώρα, αλλιώ να μου πείτε αύριο. Ωραία. Έτσι ολοκληρώνεται η συζήτηση. Σταματάμε για σήμερα μέχρι αύριο λοιπόν. Και να σας υπενθυμίσω και θα στείλω και ηλεκτρικό, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο να φέρετε τις κάρτες σας για να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Έχουμε πολλές ψηφοφορίες αύριο Γι' αυτό σας παρακαλώ φροντίστε να τις έχετε μαζί σας. Αύριο το πρωί στις 9 θα τα ξαναπούμε. Καλό βράδυ.